Κυρίες και κύριοι, θα ξαναρχίσουμε με το 17. Αναφορά 354 κάθετος 2006. Ο κύριος Μέιλο αναφέρον θα λάβει το λόγο για 5 ολόκληρα λεπτά και μετά ο κύριος Μπάκστον μαζί με τον προηγούμενο 5 λεπτά. Ο κύριος Μέιλ πρώτα. Oh. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να καταλάβει κανείς τι συμβαίνει εκεί, πρέπει να διαβάσει τα δύο βιβλία που σας έχω στείλει διαδρομή του αγωγού υγροποιημένου φυσικού αερίου που προβλέπετε δεν ταυτίζεται με τα τερματικά στα οποία πρέπει να καταλήγει. Ενώ προβλέπετε όποτε υπάρχει τέτοιο τερματικό να υπάρχει μια μελέτη που να αποδεικνύει ότι ο αγωγός ακολουθεί την λογικότερη διαδρομή. Αυτό δεν έχει γίνει. Δηλαδή τα τεστ έχουν αποτύχει, έχουν δείξει ότι δεν είναι σωστό το σχέδιο, ούτε είναι, έχουν προβλεφθεί οι, τα μέτρα ασφαλείας που έπρεπε να προβλεφθούν. Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για τους κατοίκους γύρω 25 χιλιόμετρα γύρω από τα τερματικά αυτά. Και εγώ εκεί κοντά μένω και βλέπω πόσο δυνατή είναι η καύση που γίνεται εκεί. Από την αποθήκη μέχρι το μισό δρόμο, μέχρι το σπίτι μου, όλα θα καούν άμα αρχίσει να λειτουργεί ο σταθμός αυτός. παράγονται 1,2 κιλοβάτ, δεν λέει ο μιλητής πόσο, κατά πόσον, την ώρα, το χρόνο, το μήνα, αλλά προβλέπεται για δαπάνη 5 κιλοβάτ για την ε, λειτουργία τους. Άρα δεν είναι και αποδοτικός. Προβλέπεται πριν αρχίσει να λειτουργεί το ΙΦΑ, ο σταθμός αυτός ΙΦΑ υγροποιημένου φυσικού αερίου, να έχει προβλεφθεί να αποφεύγονται προβλήματα με στατικό ηλεκτρισμό και τα λοιπά, ό,τι αντιμετωπίζουν συνήθως τα διηληστήρια, αλλά εγώ έχω δει κόσμο να καπνίζει σε απόσταση επικίνδυνη από το κέντρο. Δεν εφαρμόζονται δηλαδή οι διαδικασίες ασφαλείας είναι από τα χειρότερα μέρη για την δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου τερματικού ύφα γιατί δημιουργεί τα προβλήματα ακριβώς που προβλέπεται να αποφεύγονται από έναν τέτοιο σταθμό κυρίως προβλήματα πυρκαϊών. Τώρα γυρίζω στη δεύτερη σελίδα, δεύτερη παράγραφο. Η εγκατάσταση ενός τέτοιου σταθμού πρέπει προηγουμένως να έχει γίνει με βάση το σχεδιασμό της ασφαλούς του λειτουργίας. Αυτό δεν έχει γίνει. Και τώρα γυρίστε στη σελίδα 3, στην τρίτη παράγραφο. Είμαι εκπλήσει ότι αυτός ο σταθμός έχει θεωρηθεί κατάλληλος για τερματικό ύφα. Πάντοτε νόμιζα ανέκαθεν θεωρούσα ότι έπρεπε πρώτα να είχε γίνει μελέτη για τις προδιαγραφές ασφαλείας πριν εγκατασταθεί ένα τέτοιο σταθμός. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε καμία τέτοια μελέτη. Πολύ περίεργο αυτό, πάρα πολύ περίεργο αυτό, γι' αυτό θα γυρίσω σε λίγο. Στην τρία. Τρίτη παράγραφος. Ακόμη και τα προγράμματα αντιμετώπισης εξαιρετικών αναγκών δεν είναι τα κατάλληλα. Υπάρχουν δύο τερματικά ύφα από τις δύο πλευρές του, του λιμανιού του Milford Haven και όποτε πρέπει να σταματήσει η λειτουργία του ενός σταθμού για λόγους ασφαλείας πρέπει να σταματήσει και του άλλου. Και αυτό δεν έχει προβλεφθεί γιατί ενώ Υπάρχουν εκεί αποθηκευμένα έφλεκτα υλικά και υγρά. Αν ένα, μία από αυτές τις αποθήκες αρχίσει πυρκαγιά σε μία από αυτές τις αποθήκες, τότε μπορεί ολόκληρο το Milford Haven να κατακαεί μαζί με την περιβάλλουσα φύση. Τα δύο τερματικά ύφα είναι τελείως απαράδεκτου σχεδιασμού. Πόσο θα τα πλέον. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους θα έλεγε κανείς ότι είναι ή να, πώς να καταστρέψουν τις ζωές 20 με 50 χιλιάδων ανθρώπων. Σελίδα 5. Παρακαλώ να καταλήξετε κάποια στιγμή. Γιατί... Μάλιστα κύριε μου θα καταλήξω. Λοιπόν. Ο σταθμός αυτός λοιπόν έχει εγκατασταθεί σε λάθος μέρος και πρέπει να πάψει η λειτουργία του ή να μην αρχίσει μάλλον. Αλλιώς θα χρειαστεί να μετεγκατασταθούν, να μεταφερθούν 20 με 50 άνθρωποι γιατί θα κινδυνεύει η ζωή τους το Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορεί να δεχτεί, δεν πρέπει να δεχτεί τέτοια χαμηλές προδιαγραφές ασφαλείας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε μου. Και εγώ ευχαριστώ. Τώρα, εξ ονόματος των κατοίκων εκεί, έχουμε δύο εκπροσώπους, τον κύριο Μέιλ και τον κύριο Μπάξτον. Μαζί έχουν πέντε λεπτά, Μέιλ και Μπάξτον. Παρακαλώ να μιλήσουν ταυτόχρονα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι νομικός ε, και έχω περάσει και νομική αρρωγή ε, σε όσους ανησυχούν για τις εγκαταστάσεις κρυμμένου φυσικού αερίου και για θέματα ασφαλείας. Από τότε που και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βήθησα την Κομισιόν να κατανοήσει το ιστορικό. Έχουμε κάποιες οδηγίες ότι ε, η οδηγία 8537 δεν έχει γίνει σεβαστή. Εδώ μιλάμε για πραγματική αποτυχία να γίνει μια ποσοτική μελέτη κινδύνου και να παρουσιαστούν ποιοι είναι οι κίνδυνοι που παρουσιάζονται στον τοπικό πληθυσμό αν υπάρχει το χάρη κάποιο ατύχημα. Ο εμπειρογνώμονά μα έχει στείλει μία έκθεση που με ανάλυση αποδεικνύει τι έχει γίνει και ότι η αξιολόγηση κινδύνου δεν ε, ήταν τμήμα τη αξιολόγησης αντικτύπου, δεν έγινε καθόλου μάλιστα. Επίσης, ε, όπως ε, λέει ο κύριος Κόξ, αλλά και αναγνωρίζει και ο ίδιος ο τομέα θα μπορούσαν οι συνέπειες να είναι καταστροφικές αν συνέβαινε κάποιο ατύχημα. Κατανοώ ότι ε, οι ερωτήσεις της Κομισιόν που τέθηκαν από την Κομισιόν στην Βρετανική κυβέρνηση ε, δεν ε, επέφεραν σοβαρέ απαντήσεις και πράγματι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Άλλοι από το Milford Haven θεωρούν ότι το Κοινοβούλιο θα ενθαρρύνει την Κομισιόν να ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάσει και κάποια άλλα επιπρόσθετα μέτρα θα μπορούσαν ε, να ληφθούν αν σκεφτούμε σε πόσο κίνδυνο ε, βρίσκεται η ανθρώπινη υγεία και ότι κατάφορα παραβιάστηκε η νομοθεσία. Εκφράζουμε την εκτίμησή μας ε, απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς εδώ στις Βρυξέλλες επειδή είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση για το ζήτημα αυτό ενώ τα δικαστήρια και οι κυβερνητικές αρχές στην πατρίδα μας δεν ε, φάνηκε να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ασφάλεια των πολιτών ή για τα νομικά τους δικαιώματα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, Πρόεδρε, θα ήθελα να υποστηρίξω τον κύριο Ρόντρι Μέιλ και όλα όσα είπε και τον κύριο Ρίτσαρντ Μπάξον. Πραγματικά εκτιμούμε το πόσο ενδιαφέρεται η Κομισιόν και το Μιλό για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. όπω είπε ο κ. Μέιλ, τα ε, φορτία ΕΦΑ τώρα μετακινούνται στο Χέιντεν και έχουμε ε, και τα πρώτα φορτία. Έτσι, λοιπόν, ο κίνδυνο που είχαμε παρουσιάσει το Δεκέμβριο του 2007 ήταν τότε θεωρητική, ενώ τώρα είναι πραγματική και καθημερινά τα βιώνουν οι πολίτε της γύρω, γύρω περιοχής. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να κατανοήσετε ότι επίγουσα δράση από την Κομισιόν και ενθάρρυνση ε, αυτής της Επιτροπής μπορεί να διαδραματίσουν ε, ένα σημαντικό ρόλο για να κάνουν τη διαφορά γιατί ε, το να έχουμε μία πραγματικά περιβαλλοντική μελέτη αντικτύπου και μελέτη του κινδύνου ε, που να αξιολογεί τον κίνδυνο ή την ασφάλεια των πολιτών μπορούμε να αποδείξουμε ότι πραγματικά βρίσκεται ε, σε λάθος τοποθεσία αυτή η εγκατάσταση και Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Τώρα έχουν βιωθεί οι κίνδυνοι, μα πιέζει ο χρόνο και αν αυτή η Επιτροπή θα μπορούσε να ασκήσει πίεση, να παρατρύνει την Κομισιόν να αναλάβει δράση απέναντι στι Βρετανικέ Αρχέ, αυτό θα μα ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιατί αυτό που δεν μπορεί να διορθώσει η Επιτροπή είναι ε, αν γίνει κάποιο ατύχημα. Και έχουμε τώρα ε, και άλλο τμήμα του μέσα στο σύστημα Πάντως, ε, ουσιαστικά δεν έχει γίνει η απαραίτητη ενημέρωση, κανείς δεν έχει λάβει το φυλάδιο ακόμη και αν ε, συνέβαινε δηλαδή ένα τέτοιο ατύχημα, δεν θα ήταν δυνατό οι αρμόδιοι να λάβουν και οι θυγόμενοι να λάβουν τα μέτρα προστασίας και οι κάτοικοι δεν ξέρουν τι θα κάνουν, αν ακούσουν το συναγερμό ή αν γίνει κάποιο τύχημα. Δηλαδή δεν, έχει διανεμηθεί, δεν έχουν διαδοθεί σχετικές πληροφορίες και σε ό,τι αφορά την εταιρεία αυτοί ουσιαστικά προσπάθησαν ε, να ε, αντιταχθούν ε, και στην Κομισιόν αλλά και στην Επιτροπή για να παρουσιάσουν ένα τετελεσμένο, ένα φέτα κομπλή. Και πραγματικά εμείς εκ μέρους όλων των κατοικών που απειλούνται ζητάμε από την Επιτροπή σας να αναλάβει δράση στο θέμα αυτό και θέλουμε να υιοθετήσετε μια προσέγγιση κοινή λογικής ώστε να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Ευχαριστώ κύριο Πάτρικ Βέγκα. Um, Ευχαριστώ. Καλωσορίζω τα σχόλια που έγιναν από του αναφέροντε και τι περαιτέρω πληροφορίε ε, που έδωσαν με πρόσθετες πληροφορίες στάλησα στην Κομισιόν. Να πω ότι η Κομισιόν είναι αρμόδια για να εξετάζει μόνο τις ε, πραβίες της ε, κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην περίπτωση αυτή. Αν ε, τυχόν δηλαδή έχουν γίνει τέτοιε παρεμβάσει. Η Κομισιόν ε, δηλαδή εξετάζει τι υποχρεώσει δυνάμει τη οδηγία AEA, τη ε, οδηγία για την περιβαλλοντική ανάλυση αντικτύπου. Έχουμε και την οδηγία βέβαια για τα οικοσυστήματα, και ίσω ε, να ισχύουν εδώ, να εφαρμόζεται εδώ και οδηγία σε βέσο 2. Αλλά σήμερα εξετάζουμε την ε, οδηγία AIA και τι πιθανέ περιβιάσει. Δεν θα ήθελα να μπω σε υπερβολικέ λεπτομέρειε σε σχέση με τι υποχρεώσει που προκύπτουν από την οδηγία, αλλά να προσθέσω ότι ο στόχο είναι να διασφαλίσει ότι πριν να γίνει, ε, να δοθεί συγκατάθεση, τα έργα τα οποία μπορεί να έχουν πάρα πολύ σημαντικό αντίκτυπο πρέπει να συνοδεύονται πριν την υλοποίησή του από μελέτη αντικτύπου. Επίση υπάρχουν υποχρεώσεις δυνάμει της οδηγίας να διασφαλίσουν ότι θα ενημερωθεί κατάλληλα το κοινό και θα έχει την δυνατότητα να σχολιάσει οποιαδήποτε προτινόμενη ανάπτυξη του έργου. Αυτά είναι τα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που εξετάζουμε. Μπορώ να σημειώσω ότι η Κομισιόν ε, ήδη έχει συζητήσει αυτό το θέμα με τις ε, Βρετανικές Αρχές και βάσει των ε, πληροφοριών που μας έχει δώσει η Βρετανική Κυβέρνηση δεν είμαστε ικανοποιημένοι ότι έχουν γίνει σεβαστές διατάξεις της οδηγίας. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε δυνάμει των εξουσιών των αρμοδιοτήτων που μας δίνει η συνθήκη. κυρία Thank you, um, I just like to... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υποστηρίξω την ε, αναφορά αυτή και την αναφορά που έχει να κάνει με αυτές τις εξελίξεις. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τόσα αναφέραν οι αναφέροντες, γιατί πραγματικά το παρουσίασαν επαρκώς το θέμα και ε, έστειλαν συνεχείς επικαιροποιήσεις και σε μένα και στην Κομισιόν αλλά όλο είναι και περισσότεροι άνθρωποι και εμπειρογνώμονες, μεταλλολόγοι, μηχανικοί κτλ. αρχίζουν να εκφράζουν ανησυχίε για θέματα της ασφάλειας που έχουν να κάνουν με τον δερματικό σταθμό και τώρα πραγματικά υπάρχει φόβος ατυχήματο και είναι εντελώς απαράδεκτο οι, οι τοπικές κοινότητες να μην είναι κατάλληλα ενημερωμένε, να μην ακούνε την άποψή τους και φυσικά ε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται με το το θέμα τη ασφάλεια, γιατί δεν έχουμε καμία αξιολόγηση του κινδύνου. Εξακολουθούμε να περιμένουμε νέα στο θέμα αυτό. Επίσης, σήμερα θέλω να τονίσω το πόσο επίγουσα είναι η κατάσταση, γιατί ακούσαμε ε, ότι έχει φτάσει ε, το πρώτο πλοίο που θα ε, παραδώσει το φυσικό αέριο. Ξέρω πάντως ότι η Κομισιόν το παρακολουθεί αυτό το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πραγματική παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας και ελπίζω ότι η Κομισιόν θα κινηθεί κατεπηγόντως για το θέμα αυτό και θα ασκήσει διαδικασία επί κατά της Βρετανικής κυβέρνησης, γιατί η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα πιεστική. Υπάρχει πάρα πολύ φόβος, όπως ακούσατε και από τους αναφέροντες. Και μάλιστα υπάρχουν πολλά αποδεικτικά στοιχεία που καταδεικνύουν ε, ότι ε, όλο αυτό το εγχείρημα δεν έχει γίνει σωστά ή με ασφάλεια. Κανείς άλλος ή καμία άλλη. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά θα γράψουμε επιστολή στην Κομισιόν. Ο εκπρόσωπός της άκουσε όσα είπατε και γνωρίζει τις ανησυχίες και αμφιβολίες σας και θέλουμε λοιπόν να απευθύνουμε επιστολή στην Κομισιόν όπου να της ζητάμε να διασφαλίσει το σεβασμό με την, στο τερματικό εκείνο με την ενωσιακή νομοθεσία και με την ασφάλεια των κατοίκων, με την προδιαγραφές ασφαλείας των κατοίκων. Την κρατάμε ανοιχτή λοιπόν την υπόθεση. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα το... Εάν δεν απατώμε το... 18. Το Ξαναλέω, κυρίες και κύριοι, δίλεπτο διάλειμμα. Ο Δαβίδ Λό θα έρθει σε επαφή με τους αναφέροντες εκεί πέρα, μήπως κάνουν καμία πρόταση. guys, the European Commission listened to their political and addressed letters to the Commission so you asking them to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

Το επόμενο σημείο είναι το 18 αναφορά 1077 2008 και ποιος θα εκπροσωπεί τους αναφέρονται, ποιος ήταν της κυρίας Ρομπέρ, της κυρίας Μπουρνιόν, του κυρίου Ρομπέρ, μήπως είναι κανείς από αυτούς παρόν. Α, ωραία, έχει πέντε λεπτά τότε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρόμοιο θέμα ή με το προηγούμενο. Είναι άλλη περιφέρεια βέβαια, άλλη τοποθεσία. Αλλά αφορά επίσης ένα σχέδιο που ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί. Αντίθετα από την προηγούμενη περίπτωση είναι σχέδιο Ολλανδοαμερικανικό που το έχει αναλάβει η Κάτρ η ίδια με το Milford Haven και το συνταξιοδοτικό ταμείο Carlisle Riverstone στο οποίο ανήκει και η οικογένεια Bush. Είναι πραγματικά κυκλόπιο έργο τύπου σε Βέσο 2 και θέτει σε κίνδυνο δύο τουλάχιστον καταπράσινες περιοχές της Γαλλίας. Εμείς είμαστε μια ομάδα πολιτών που γνωρίζουν τα πράγματα και θα θέλαμε να γνωρίζετε κι εσείς ότι αυτό το πρόγραμμα αποθήκευσης ε, μεθανίου αποτελείται από τρία ρεζερβουάρ 85 μέτρων διαμέτρου και 47 μέτρων ύψους ο όγκος που μπορεί να κρατηθεί εκεί είναι 165.000 κυβικά μέτρα, δηλαδή συνολικά 495.000 κυβικά μέτρα. Είναι τεράστιος όγκος. Εκτός από αυτή την αποθήκευση υπάρχουν μία ομάδα επαναεριοποίησης, μία ομάδα που προσθέτουν τοξικές ουσίες για να έχει μυρωδιά το αέριο, το οποίο είναι τύπου RSH, ένα κέντρο που μεταφέρει το προϊόν αλλού και όλα αυτά αντιπροσωπεύουν σημαντικούς κινδύνους και γι' αυτό το λόγο ο Ευρωπαίος Νομοθέτης τέτοιου είδους εγκαταστάσεις ονομάζει τύπου σε βέσο 2 ανωτά του επίπεδου κινδύνου. Η Γαλλία με μεγάλο κόπο κατόρθωσε να καθορίσει ορισμένες παραθαλάσσιες ζώνες της ως διατηρητές στο Natura 2000. Ε, όμως μέσα στη μέση της ζώνης αυτής Natura 2000 αυτό το σχέδιο πήγασος προβλέπεται να δημιουργηθεί. Κατά παραβίαση της ταξινόμησης Natura 2000 και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας του Περιβάλλοντος όπως οι οδηγίες για τους βιότοπους και για τους ε, ορνηθότοπους. Το δέλτα του Ζιρόντ καθώς και το τέλμα Μπέκ Νταμπές έχουν ταξινομηθεί ως σημαντικές, σημαντικές περιφέρειες της ε, βιογεωγραφικής περιφέρειας εκείνη σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Κομισιόν. Εκτός αυτού η γεωλογική ποικιλομορφία του υπεδάφους εκεί είναι τελείως ιδιαίτερη. Είναι πολύ ευαίσθητο υπέδαφος και υπάρχουν εκεί εναποθέσεις ασβεστίου που δημιουργήθηκαν ε, στην προϊστορική εποχή από εναποθέσεις των ποταμών καθώς και κατάλοιπα φυτών, τύρφης κλπ. Αυτά όλα πολύ εύκολα μπορούν να υποστούν διάβρωση καθώς και τις επιπτώσεις ε, καιρικών φαινομένων καθώς και της παλήριας. Επίσης έχουν την ιδιότητα να καθιστούν ακόμη σοβαρότερη οποιαδήποτε σεισμική δόνηση το 1999 είδαμε ότι η ξαφνική άνοδος του επίπεδου της θάλασσας δημιούργησε φαινόμενα τύπου τσουνάμι. Το γεωλογικό παρελθόν της περιοχής είναι επίσης ιδιαίτερο. Η Ιβυρική πλάκα συγκρούστηκε με την Ευρωπαϊκή και έτσι δημιουργήθηκε η περιοχή με αποτέλεσμα τη δημιουργία των Πυρηναίων. Έτσι η αριστερή και η δεξιά όχθη της Ζηρών διαφοροποιήθηκαν τελείως. Από τη μία πλευρά η πλάκα ανεβαίνει, από την άλλη κατεβαίνει. Και στις εκβολές του ποταμού το νησί Ολερών είναι σεισμογενές. Παρακαλώ να καταλήξετε. Ε, πώς να καταλήξω κύριε Πρόεδρε αφού έχω ακόμα τρεις σελίδες. Ήδη ξόδεψα πέντε λεπτά. Να συνεχίσω. Α, τότε καλά. Πού ε, ήμουνα, στις εκβολές του. Α, όχι, την τελευταία, η τελευταία σοβαρή κρίση της νήσου της Ολερών έγινε το Σεπτέμβριο του 1972. Αλλά υπήρξαν κι άλλες παλαιότερες κρίσεις σημαντικές. Ο μεγάλος κατακλυσμός του 580, οι σεισμοί του 1427 και 1428 καθώς και άλλες μικρότερες κρίσεις, άλλα που συνεχίζονται. Αυτές οι Αυτά τα σεισμολογικά φαινόμενα μπορούν να δημιουργήσουν τσουνάμια στην περιοχή Μεντόκ. Το Φεβρουάριο του 1924 δημιουργήθηκε ένα παλιροϊκό κύμα πολύ σημαντικό για την περιοχή και οι απόκριμνες ακτές της περιφέρειας εκείνης που δημιουργήθηκαν από τις αναποθέσεις των ποταμών μπορούν να δημιουργήσουν ακόμη σοβαρότερα προβλήματα στο μέλλον εάν υπάρξει κάποιο τέτοιο καιρικό γεωλογικό φαινόμενο. Το Δέλτα μειώνει το εύρος του και γι' αυτό μπορεί να αυξηθεί η δύναμη των παλιριών που, και των παλιριωικών κυμάτων που μπορεί να δημιουργηθούν εκεί. Έχουν ληφθεί βέβαια κάποια μέτρα, έχει χτιστεί κάποιο αντέρισμα και τεχνητή βράχη, αλλά αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ε, θύελα ισχύω 4 όπως το 99. Και αν μεταξύ όλων αυτών δημιουργηθεί και ένα κέντρο αναποθηκεύσης μεθανίου, τι θα γίνει αν γίνει κάτι σαν το 580 ή το 1427-28, θα υπάρξει έκρηξη του μεθανίου και θα καταστραφούν έτσι και οι υπόλοιπε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Βέβαια έχουμε μιλήσει μόνο για φυσικά φαινόμενα, αλλά αυτά είναι ικανά να μας σβήσουν από το χάρτη. Δεν αποκλείεται να υπάρξει ένα τέτοιο ατύχημα με το μεθάνιο αν εγκατασταθεί. Γιατί ο κύριος λόγος για τον οποίο παρέμεινε σε αγρίαν κατάσταση αυτό το δέλτα του ποταμού είναι ότι δεν υπήρχαν τόσο πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Παλιά ήταν μάλιστα λιμέρι πειρατών. Σας παρακαλώ, ευχαριστούμε κυρία μου, ευχαριστούμε. Καταλάβαμε. Όχι, τελειώσατε ήδη. Μα δεν καταλαβαίνω πολωνικά, γι' αυτό δεν κατάλαβα. Είπατε να τελειώνω. Ήδη 8 λεπτά πήρατε, κύριε, 8 λεπτά. Α, τότε καλά. Δεν δουλεύει το μικρόφωνο, γι' αυτό ακούγομαι. Λοιπόν. το πευκόδασος εκεί θα εξετίθετο σε ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες αν συνέβαινε κάποιο τέτοιο ατύχημα. Σε αυτή την προεκλογική περίοδο δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες πώς μπορεί η νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος να μην εφαρμόζεται. Αυτό δίνει πρόσθετα επιχειρήματα στους εχθρούς της Ευρώπης που έλεγε ότι θα τους προστατεύει στην καθημερινή του ζωή. Για την ιστορία, τη γεωλογική ιστορία της περιοχής θα σας παραπέμψω. Σας ευχαριστώ πολύ, τελειώσατε. Ο κύριος Ρομπέρ ή η κυρία Ρομπέρ. Ε, Κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής Αναφορών, σας ευχαριστώ θερμά που εκτιμήσατε τη βαρύτητα του θέματος που έχουμε θέσει για το θέμα της αποθήκευσης μέσα υγροποιημένου φυσικού αερίου στον, στις του Ζιγόντ. Δεν θα σχολιάσω περαιτέρω τις ειδικές λεπτομέρειες της αναφοράς, έχουν ήδη αναλυθεί. Εγώ θα ήθελα απλώς να αναφερθώ στο νομικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο του θέματος αυτού, στην συγκεκριμένη κοινότητα. Η διαχείριση της γης είναι σημαντικό θέμα. Έχουν ε, γίνει το ένα πρόβλημα που τίθεται είναι ότι αυτή η εγκατάσταση θα ε, κατασκευαστεί σε περιοχή Natura 2000. Είναι λοιπόν ένα ερώτημα, ποια δικαιοδοσία, ποια αρχή είναι αρμόδια για να πάρει μια τέτοια απόφαση. Υπάρχουν ε, οι τοπικές αρχές οι οποίες, ε, στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει η διαχείριση αυτής της περιοχής. Ένα ερώτημα λοιπόν που θέτεται είναι ποια είναι η θέση της εταιρεία που έχει αναλάβει αυτό το έργο έναντι των αρχών αυτών. Υπάρχουν θέματα και όσον αφορά την, το εργασιακό καθεστώς και τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα των φορολογούμενων. Μας ενδιαφέρει. Τίθενται λοιπόν θέματα Συνειδητοποιείτε λοιπόν ότι η απόφαση που θα λάβετε όσον αφορά αυτή την αναφορά για την κατασκευή αυτού του τεράστιου έργου που αποτελεί, σε μια περιοχή που αποτελεί περιοχή φυσικού κάλους και πόλο έλξη τουριστών είναι σημαντική. Αν δεν υποστηρίξετε αυτό το, τη, θέση μας, τίθεται το ερώτημα τι νόημα έχουν οι περιοχές Natura 2000 και ποια είναι η προοπτική που, δίνουμε στον πλανήτη. Ευχαριστώ. Bardzo dziękuję. Pani Josiane Bardzo proszę. Josiane Ευχαριστώ πολύ την Κομισιόν που τοποθετήθηκε θετικά σε σχέση με το παραδεκτό της αναφοράς ε, που θα εξετάσετε. Ευχαριστώ λοιπόν την Επιτροπή. Εγώ είμαι τακτικό μέλος της ΕΛΠΕΟ, του Ιδρύματος Νικολάηλο και προέρχομαι από το Διοικητικό Συμβούλιο της Καριμά, η οποία διαχειρίζεται τον υγρότοπο στο Βερντόν Σιμέρ ε, και είναι πολύ φιλική κατάσταση γιατί ανήκει είτε στην κοινότητα είτε στο Γενικό Συμβούλιο ε, είτε στο θαλάσσιο λιμένο του Μπορντό. Ε, λοιπόν, για το πρόβλημα που μας απασχολεί εδώ, ευχαριστώ την Κομισιόν προσωπικά αλλά και εξ ονόματος όλων όσων εργάστηκαν για την υποβολή αυτής της αναφοράς μια τόσο σημαντική ένωση λόγω του αριθμού των μελών τη ή λόγω του αντικτύπου των δράσεών τη δεν θα μπορούσε να απαντήσει ε, σε όλες αυτές τι προκλήσεις ε, αυτών των ε, τόσων πολλών ανθρώπων που αντιτίθενται στο μεθάνιο. Αυτή η αναφορά γεννήθηκε λοιπόν εκτός τη Ένωση, κατά τη διάρκεια μια δημόσια συζήτηση, ιστορικού χαρακτήρα. Ουσιαστικά αποτελεί φωτογραφία ε, των ανησυχιών ε, ενός ε, πληθυσμού των μονίμων κατοίκων και των κατοίκων που έρχονται να περάσουν τις διακοπές τους. Για να ξεκινήσω, όταν μιλάμε για την Κατριγκάς, είναι ο κύριος του έργου. Θέλουμε να αναφέρουμε τον ιδιαίτερα σταθή χαρακτήρα αυτών των χρηματοπιστωτικών ομίλων και επίσης ε, θέλουμε να πούμε ότι δεν ενδιαφερόνται καθόλου για την αηφόρο ανάπτυξη σήμερα. Ε, αποκαλούνται ουσιαστικά κυρίως το έργο, αλλά αύριο που είναι η δημόσια συζήτηση δεν, δεν κατόρθωσε να πείσει για το σημείο αυτό, παρόλο που το θέμα τέθηκε επανειλημμένα. Επίσης, ανανεώνω τα ερωτηματικά σε ό,τι αφορούν αυτό τον αγωγό αερίου, γιατί ε, στο φάκελο του τερματικού του μεθανίου δεν έχει συμπεριληφθεί αφού τα δύο αυτά έργα ε, δεν ε, διαιρούνται μεταξύ τους. Ε, όλοι το υπογραμμίζουν. Πολλές φορές έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει έλλειψη πληροφοριών από τις δημόσιες αρχές. Η σύμβαση πάντοτε, πρέπει να γίνεται, πάντοτε έγινε σεβαστή και εγώ ίδια έθεσα αυτό το ερώτημα και από τον Ομάρχη έλαβα την απάντηση ότι το κράτος και οι υπηρεσίες τους δεν μπορούσαν να μας ε, ενημερώσουν αν δεν είχε ολοκληρωθεί το έργο ή αν η κοινώση θα γινόταν μέσω του τύπου. Η επικοινωνία θα γινόταν μέσω του τύπου ενώ ταυτόχρονα η Κάτερ ε, ουσιαστικά έστελνε ε, μία πλακέτα σε όλους τους κατοικούς ε, του Μεντόκ. Πολύ μεγάλη αντίθεση εδώ. Ε, να σας πω ότι στέλνω στην γραμματεία κάποια έγγραφα που μπορεί να έχουν στην κατοχή τους στη συνέχεια όλα τα μέλη. Σε μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις εργασία η οι 11 κοινότητες εξέτασαν το σχέδιο της βιώσιμης ανάπτυξης εξή ε, και τοποθετήθηκαν κατά οποιοδήποτε έργο που παρουσίαζει κίνδυνο είτε για τη φύση είτε από τεχνολογική σκοπιά. Ε, ε, μιλάμε εδώ, παραδείγματο χάρη, για διάβρωση τη αρχή για ορισμένου τομεί, που είναι δύσκολο να του προστατεύσουμε. Μιλάμε, εδώ έχουμε μία μάχη αδιάκοπη κατά των στοιχείων και φυσικά οι συνέπειες της αλλαγής του κλίματος ε, τίποτα δεν θα λύσουν. Ε, ε, βλέπουμε πόσα πουλιά πεθαίνουν στις παραλίες και βλέπουμε πόσες είναι οι συνέπειες στην Πανίδα και στη Φλωρίδα. Μην ξεχνάτε εδώ ότι μιλάμε και για επιπτώσεις στο πιο μεγάλο, σε ένα από τα πιο μεγάλα δάση της Ευρώπης. Επίσης ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη τι θα γίνει με ε, την ναυσιπλοεία ε, στην περίπτωση που υλοποιηθεί το έργο της Πεγκάς. Οι σεισμικοί κίνδυνοι δεν έχουν ληφθεί υπόψη και ουσιαστικά δεν ξεκαθαρίζεται γιατί έχει επιλεχθεί αυτό αυτή η τοποθεσία ουσιαστικά οι σεισμικοί κίνδυνοι θα αποτελούσαν πολύ, μεγάλους, πολύ μεγάλη απειλή. Όταν ε, οι τεχνολογικοί κίνδυνοι παρουσιάστηκαν ε, στο Κογκρέσο, στο Σουλάξ μέρα από τις αρμόδιες αρχές, ε, ουσιαστικά έμοιαζε με μια τραγική, είχε μια τραγική εξέλιξη, γιατί ποιος θα δεχόταν τελικά να έχει στην πόρτα του ένα τέτοιο κίνδυνο. Και το εργοστάσιο της Μπλάγη ουσιαστικά δεν αρκούσε για να έχουμε ε, τόσες επικίνδυνες ενέργειες. Ήταν λογικό να σκεφτούμε ότι θα έχουν οι πολίτες ένα τέτοιο κίνδυνο στην πόρτα τους. Αν μπορείτε να κλείσετε, λέει ο Πρόεδρος. Μάλιστα. Κλείνω. Υπάρχουν ε, κάποια είδη που απειλούνται, το είπαμε αυτό, ε, παραδείγματο χάρη το, τα χέλια, ε, έχουμε ε, στην περιοχή αυτή ε, και ε, ήδη αεροπλάν, αεροσκάφη που περνούν και ουσιαστικά αυτό έχει επιπτώσει στα μεταναστευτικά πτηνά. Επίσης έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τη γεωργία, με την δεδοκολιέργεια και αυτό θα έχει συνέπεια στις δραστηριότητές τους και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι εμείς που κατοικούμε στο Δέλτα στην εκβολή του Πετικού είμαστε θύματα όπως και όλοι οι κάτοικοι των Δέλτα των ε, ποταμών του κόσμου. Μπορείτε να δείτε τι συνέβη και στο Κολοράντο ε, έτσι λοιπόν, ε, θέλω, θέλω να πω ότι η Ένωση επειδή ενδιαφέρεται για τη δική μας ε, περιφέρεια θα έπρεπε να προσπαθήσει να την προστατεύσει. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Εμείς έχουμε λάβει το υλικό από εσά, τα σχετικά έγγραφα. Και φυσικά το μελετήσαμε. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον Πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Αντουάν Ποντούς. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτέ, είμαι εκπρόσωπος μιας οργάνωσης που καταπολεμάει το σχέδιο αυτό και που δημιουργήθηκε πριν από περίπου δύο χρόνια, μόλις μάθαμε τα σχέδια αυτά. ακούσατε αυτά που είπαν οι φίλοι μου που κατέθεσαν την ε, αναφορά. Θα ήθελα εγώ να προσθέσω ότι ως επένδυση το σχέδιο αυτό αντιπροσωπεύει ένα εκατομμύριο ευρώ μαζί με τη δημιουργία του αεριαγωγού στο τελευταίο φυσικό ποτάμιο δέλτα της Ευρώπης. Η τοποθεσία είναι πολύ σημαντική από άποψη βιοπικιλότητας γιατί εκεί ζουν πάρα πολλά προστατευόμενα είδη και βρίσκεται δίπλα ή στο κέντρο μιας περιοχής αναγνωρισμένης από το Natura 2000 και που προστατεύονται από την οδηγία των πετινών και των βιοτόπων καθώς και της πανίδος και χλωρίδος. Η... Το σχέδιο αυτό, το πρόγραμμα αυτό θα καταστρέψει τη βιοποικιλότητα αυτήν στην περιοχή εκείνη του βορείου Μεντόκ. Ποια, ποιο είναι το ενδιαφέρον για το κοινό. Αν, είχε, αν υπήρχε τέτοιο ενδιαφέρον θα λέγαμε, ε, τι ενδιαφέρον έχει το βασχέδιο μάλλον, αν είχε κάποιο, κάποια τέτοια σημασία θα λέγαμε δεν πειράζει η οικολογική ζημία. Αλλά οι μελέτες δείχνουν ότι το 2015 η Γαλλία θα έχει υπερβολικές ποσότητες αποθηκευμένου αερίου και η Ευρώπη επίσης φυσικού αερίου υγροποιημένου. Ας μην σας δώσω αριθμούς, αλλά υπάρχουν όμως στα έγγραφα που θα σας παραδώσω. Το σχέδιο λοιπόν αυτό αντιπροσωπεύει πολύ σημαντικό κίνδυνο για το χωριό που βρίσκεται 100 250 μέτρα από το κέντρο αυτό και παρά τι διαμαρτυρίες που ακούστηκαν, το μόνο που έκανε ο επενδυτή είναι να καταθέσει ένα νέο σχέδιο ανάλογο με το παλαιότερο. Υπάρχει και ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που θα σας δώσω, καθώς και ένα άλλο που αναφέρει πού βρίσκονται ακριβώς τα πράγματα. Η οργάνωσή μας λοιπόν καλεί τους ευρωβουλευτές αν θέλουν να έρθουν να δουν με τα μάτια τους πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και ποιο Ποιε θα είναι οι κοινωνικο οικονομικέ αλλά και περιβαλλοντολογικές ζημίε, αν τελικά πραγματοποιηθεί αυτό το σχέδιο της Ολλανδοαμερικανική Εταιρεία Κάτρα Γκάζ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Didier Καντά που είναι μέλος της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Κύριε Πρόεδρε, ως Γάλλος βουλευτής θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και εσάς και τα μέλη της Επιτροπής σας για την πρόσκλησή σας γιατί πράγματι είναι χρήσιμο δημοκρατικά να ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Τιούτων. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ. Μετά από αυτά που ακούσαμε από, τους, ε, από τις οργανώσεις που τίθενται κατά του σχεδίου αυτού. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας πω για ποιους λόγους ο, οι κάτοικοι της περιοχής εκείνη σχεδόν ομόφωνα κατά του σχεδίου αυτού για την εναποθήκευση μεθανίου στο τελευταίο αυτό φυσικό ποτάμιο δέλτα της Ευρώπης. Νομίζω ότι θα καταλάβετε ότι είναι τριπλά παράλογο ενεργειακά, οικολογικά και οικονομικά το σχέδιο αυτό και ότι επομένως πρέπει ως το δυνατόν συντομότερα να καταργηθεί, να μην εφαρμοστεί. Είναι παράλογο ενεργειακά καταρχήν, διότι η Γαλλία ήδη έχει υπερβολικά μεγάλες ποσότητες αποθηκευμένου υγροποιημένου αερίου ο πρόεδρος των Γαλλικών Λιμένων Μισελ Κεμπέρ δήλωσε τελευταία ότι με την αύξηση της δυνατότητας αναποθήκευσης που υπάρχει στη Βρετάνη θα έχουμε τέσσερις φορές παραπάνω αποθήκευση από όσοι χρειαζόμαστε. Και πρόσθεσε ότι δεν είναι καθόλου απαραίτητο να γίνει μια νέα εγκατάσταση αποθήκευσης υγροποιημένου μεθανίου, ότι πρόκειται για κερδοσκοπία αφού υπάρχουν ήδη τα άλλα στη Δανκέρκη και τη Χάβρη. Επομένως, είναι τελείως παράλογο εφόσον μάλιστα στην Ισπανία προς τον Μπιλμπάο και αλλού υπάρχουν ήδη τέτοιες αποθήκες. Είναι επίσης παράλογο οικονομικά διότι η δημιουργοί του σχεδίου λένε ότι θα υπάρχουν πολύ μεγάλα οικονομικά ωφέλη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό όμως θα είναι ελάχιστο αν το συγκρίνουμε με την καταστροφή που θα υποστεί η τουριστική βιομηχανία εκεί. Πράγματι, αν αυτό το σχέδιο πραγματοποιηθεί, τότε σύμφωνα με τους υπολογισμούς μείωσης του τουρισμού, μεταξύ 400 και 1000 θέσεων εργασίας θα καταστραφούν εκεί και θα συμπαρομαρτούν τα βέβαια. Επίσης, υπολογίζεται σε 30 με 90 εκατομμύρια ευρώ ο οικονομικός γύρος ε, που θα δημιουργηθεί, ενώ ο τουρισμός είναι πολλαπλής τέτοια τάξης γύρω στα 600 εκατομμύρια. Επίσης είναι παράλογο και οικολογικά, διότι οι επιπτώσεις του θα είναι καταστροφικές για τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον, βιοποικιλότητα που είναι ιδιαίτερα πλούσια εκεί και για τη χλωρίδα και για την πανίδα. Μια τέτοια εγκατάσταση θα δημιουργήσει οπτική μεταξύ άλλων ε, ε, μόλυνση και προστίθενται οι κίνδυνοι για την αυσιπλοεία διότι τα πλοία που μεταφέρουν μεθάνιο που είναι πάνω από 400 μέτρα μήκους ε, πρέπει να έρχονται εκεί από ένα κανάλι που είναι ιδιαίτερα ρηχό για τέτοια πλοία θα καταστραφεί ο σταθμός του κλαμπ τερανέ Παλμύρα καθώς και άλλα θέρετρα. Τα πλοία λοιπόν αυτά εκτός των άλλων θα εναποθέτουν εκεί και βαρέα μέταλλα που θα βλάψουν ιδιαίτερα και την οστρεοκαλλιέργεια και την αλληλεία εκεί. Η περιοχή εκείνη είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τη Γαλλία και για την Ευρώπη περιβαλλοντολογικά. Γι' αυτό είμαστε πεπισμένοι ότι υπάρχουν άλλες δυνατότητες ανάπτυξης για το αυτόνομο λιμάνι του Μπορντό, πολύ λιγότερο βλαπτικές για το περιβάλλον από ό,τι το σχέδιο αυτό. Και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που η γαλλική κυβέρνηση στις 20 Ιουνίου 2008 απάντησε θετικά στο αίτημά μου δημιουργίας μη προστατευμένης θαλάσσιας ζώνης εκεί γύρω και στην κοντερή Ρουαγιάλ του Ροσφόρ ήδη δημιουργήθηκαν γραφεία για τη διαχείριση της ζώνης εκείνης και για την προστασία της ζώνης ολόκληρης. Η γαλλική λοιπόν κυβέρνηση στα πλαίσια της οικολογικής διάσκεψης Γκρενέλ είχε προβλέψει ολόκληρη δέσμη μέτρων για αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών όπου αναγνωριζόταν ότι η περιοχή εκείνη, ο μεγαλύτερο ποτάμιο δέλτα της Ευρώπης είναι πολύ σημαντικός παράγοντας τουρισμού. Η προστασία της χλωρίδας, της πανίδας και των πετινών εκεί είναι επίσης κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και μπορεί κανείς να αναρωτηθεί τι σημασία θα είχε η δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου μπροστά σε τέτοιες αρνητικές οικολογικές συνέπειες. Κυρίες και κύριοι βουλευτέ, η τοπική μας οικονομία δεν θα μπορέσει να αντέξει για πολύ ακόμα αυτή τη δαμόκλεια σπάθη που τίθεται πάνω από το κεφάλι της. Υπάρχει εδώ κάτι το οποίο ξεπερνάει κατά πολύ την τοπική μονοδιάσταση. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω την κινητοποίηση και, την κινητοποίησή σας ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την περιοχή εκείνη και καλώ μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής σας να έρθει να επισκεφθεί εκεί το μέρος για να δείτε τι συμβαίνει. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα εδώ να θυμίσω τις ε, τους διάφορους κανονισμούς που ισχύουν. Υπάρχει η οδηγία για τους οικοτόπους και τα πτηνά Κάθε έργο που αφορά τη διαχείριση του, της περιοχής αυτής πρέπει να αποτελεί αντικείμενο κατάλληλης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελέτης για τη διατήρηση του φυσικού οικοσυστήματος. Πρέπει να δοθεί σχετική έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να μην πληγεί η ακεραιότητα του οικοσυστήματος. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία για τους οικοτόπους, αν η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει καταλήξει σε, αρνητικό, σε αρνητική εισήγηση, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο, στο κοινό, στο δημόσιο συμφέρον και να ληφθούν όλα τα μέτρα, όλα τα αντισταθμιστικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η εναρμόνιση με, τη, με τις αρχές που διέπουν τις περιοχές Natura 2000. Όσον αφορά τώρα την αποθήκευση αερίου και ανάλογες εγκαταστάσεις, πρέπει και πάλι να γίνεται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υπάρχει σχετική νομοθεσία για, που αφορά όλα τα έργα ιδιωτικής ή κρατικής πρωτοβουλίας. Υπάρχει επίσης οδηγία σχετικά με την πρόληψη της ρήπανσης και η οδηγία για, την, ε, για το περιορισμό ορισμένων ε, ε, ρήπων στην ατμόσφαιρα από μονάδες καύσης. Η περιοχή του, η περιφέρεια Ζιρόντ έκανε, έχει διαπιστώσει κενά στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχει εκπονηθεί μια σχετική έκθεση και αυτή τη στιγμή δεν διαπιστώνεται παραβίαση της ε, οδηγίας για τα πτηνά και σύμφωνα με και η Επιτροπή θα παραμείνει, ε, θα εξακολουθήσει να ασχολείται με το θέμα, να ελέγχει κατά πόσο τηρούνται οι οδηγίες και η νομοθεσία για τις περιοχές Natura 2000. Η Κομισιόν επίσης θα έρθει σε επαφή με τις γαλλικές αρχές ώστε να, ελαχιστο... να φροντίσει για την ελαχιστοποίηση του αντικτύπου στην περιοχή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ονέστ. Σας ευχαριστώ. δεν είμαι υποψήφιος για τις εκλογές του Ιουνίου. Δεν, κάνω κανενός είδους πολιτική εκστρατεία. Ο λόγος που είμαι εδώ, αυτό που θέλω να πω είναι να δηλώσω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι απολύτως σοβαροί. Εγγυώμαι γι' αυτό προσωπικά. Είναι σπάνιο φαινόμενο να βλέπουμε τέτοια σύμπνοια μεταξύ πολιτών και εκπροσώπων τους και αιών τους. Είμαστε αντιμέτωποι με ανθρώπους που ο μόνος λόγος που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και μιλάω για την εταιρεία είναι το κέρδος. Ο μόνος λόγος, το μόνο, η μόνη τους έγνοια είναι αυτή και πολύ, την επόμενη φορά θα σε κάποια άλλη ανάλογη περιοχή και πάλι με στόχο το κέρδος. Μιλούμε για περιοχή Natura 2000, μέρος της οποίας είναι και θαλάσσιο οικοσύστημα. Από τεχνολογικής άποψης μιλούμε για ένα έργο εξαιρετικά ευαίσθητο. Είναι ένας αγωγός αερίου. ο οποίος θα έχει τη δυναμικότητα τετραπλάσια της απαιτούμενη για την κάλυψη των αναγκών της χώρας. Κλήθηκα ενώπιον του δικαστηρίου για να εκθέσω την άποψή μου. Εδώ και πολλά χρόνια επιμένουν ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι, ότι γίνονται όλοι οι έλεγχοι. Υπήρξαν ωστόσο, εγώ προσωπικά έχω βιώσει ατυχήματα με θύματα, καταστροφή του περιβάλλοντος και δεν θα ήθελα να δω το ίδιο πράγμα να συμβαίνει και σε αυτή την περιοχή. Πρόκειται για μια δαμόκλειο σπάθη που απειλεί όλους τους κατοίκους αυτής της περιοχής και είναι σπάνια η ευκαιρία που δίνεται σε μέλη, σε βουλευτές να αποφασίσουν τη μοίρα μιας περιοχής, αν θα συνεχίσει να υπάρχει ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Χαμερστάιν, παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας ακόμη περίπτωσης ε, που ε, πραγματικά ε, βλέπουμε να απειλείται ένα πάρα πολύ, μια πάρα πολύ σημαντική τοποθεσία εκβολής ενώ μου, εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω την Κομισιόν ε, να ε, δράσει πιο γρήγορα για την υιοθέτηση του σχεδίου για την προστασία θαλάσσιων περιοχών ε, και να προωθήσει το πώς γίνεται η στρατηγική ανάλυση σε σχέση με τις ορευτικές συνέπειες σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο που έχουν οι πετρελαγωγοί και τα ηλεκτρικά δίκτυα και επίσης ε, να τοποθετηθεί και ε, σε ό,τι αφορά την έλλειψη εναλλακτικών που να έχουν μελετηθεί. Εγώ πάντοτε πραγματικά ρωτιέμαι γιατί δεν χρησιμοποιούνται ήδη βιομηχανικά βεβαρημένες τοποθεσίες, γιατί πάντοτε επιλέγουν παρθένες περιοχές για να φτιάξουν αυτά τα έργα. Έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει να δούμε τη δυνατότητα εναλλακτικών αλλά και την εναλλακτική, τη μηδενική δηλαδή να μην γίνει καθόλου ένα τέτοιο έργο. Ευχαριστώ. Η κυρία προστασία των περιβάλλοντων αλλά και την ασφάλεια του τοπικού πληθυσμού. Έτσι λοιπόν ε, θα ήθελα να ενθαρρύνω την Επιτροπή να συνεχίσει, να δώσει συνέχεια σε αυτή την αναφορά. Ευχαριστώ. Κύριος Κάσμαν, καταρχήν ε, να σας ε, πω θα, σας, θα μας λείψετε Ερνέστο στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά που έχετε κάνει σε αυτό το κοινοβούλιο εκπροσωπώντας την περιφερειά σας και τη χώρα σας. Νομίζω ότι αυτή η αναφορά θέτει πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Έχουμε κοινωτική νομοθεσία η οποία δεν γίνεται σεβαστή. Ε, εγώ λοιπόν θέλω να ζητήσω από την Κομισιό να μας δώσει περαιτέρω πληροφορίες και υποστηρίζω ένθερμα τις τρεις αναφορές που έχουμε ενώπιόν μας. Αναμένω λοιπόν να ακούσω ποιες θα είναι οι έρευνες στι οποίες θα προβεί η Κομισιόν εκ μέρους μας. Κυρίες και κύριοι, είχαμε μία μακροσκελή συζήτηση για το θέμα αυτό. είναι η συνήθειά μας να ξαναδίνουμε το λόγο στους συντάκτες των αναφορών, αλλά είναι δύσκολο τώρα να δώσουμε το λόγο σε όλους όσους είναι παρόντες. Νομίζω λοιπόν ότι το καλύτερο θα ήταν να γίνει μια σύνοψη από τον κύριο Καντέν. Σας παρακαλώ, μπορείτε να συνοψίσετε τη συζήτηση με δύο λόγια, μαζί και μόνο αυτά που ακούσαμε από την Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι ακούσατε όλο το βεληνικές των επιχειρημάτων ε, κατά αυτού του έργου από τη δική μας σκοπιά επαναλαμβάνω ότι δεν έχει νόημα, δεν έχει κανένα νόημα από ενεργητική σκοπιά γιατί ήδη έχουμε αποδείξει ότι έχουμε υπερδυναμικότητα αποθήκευση στην Γαλλία με τα έργα τα οποία έχουμε κατά νου, όχι μόνο για την Γαλλία αλλά και για την Ισπανία. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει νόημα από ενεργητική σκοπιά ούτε από οικονομική σκοπιά γιατί γιατί οι θετικέ συνέπειε ε, θα ήταν πολύ μικρότερε από τι αρνητικέ ε, σε ό,τι αφορά τι επιπτώσει ε, στον τουρισμό αλλά και τι πρωτογενεί δραστηριότητε, αλλήλια, το καλλιέργεια κτλ. Και από οικολογική σκοπιά να αναφέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Ήμουν λίγο βουλευτή στην περιοχή και πραγματικά έχουμε στο παρελθόν και τι τελευταίε δεκαετίε αλλά και του περισμένου αιώνε, ιδιαίτερη σεισμική δραστηριότητα. Βλέπετε λοιπόν όλου αυτού του κίνδυνου. Σα παρακαλώ, μην πιστέψετε ότι είμαστε ε, εδώ υπέρ του σκοταδισμού στη Γαλλία. Έχουμε άλλες ε, τοποθεσίες στην ακτή που μπορούν να ε, υποδεκτούν τέτοιες παραδείγματο χάρη εγκαταστάσεις. Έχουμε στην Βρετάνη τέτοιες περιοχέ και έχουμε και το project του Ντανκέρ. Έχουμε δηλαδή εκβολές που μπορούν να εξυπηρετήσουν τέτοια βιομηχανικά σχέδια ενώ έχουμε άλλες περιοχές όπω είναι οι Ζιρόντε που ε, έχουν ουσιαστικά έναν οικολογικό χαρακτήρα. Σας είπα ότι είναι ο πιο μεγάλος ε, το πιο μεγάλο ε, δέλτα στην Ευρώπη. Και πώς θέλουμε να περάσει επίσης ένας αγωγός αερίου μέσα από όλους τους αμπελώνες του Μπορντό. Δηλαδή θα περνούσε από κάπου μεταξύ του Ρεγιό και του Σαζόρ Δεν νομίζω ότι ε, θα το εκτιμούσαν αυτό οι αγρότες. Έτσι λοιπόν ε, είστε ενώπιον ανάληψης οικολογικής ευθύνη και ιστορικής θα έλεγα, χωρίς να φοβάμαι τις λέξεις. Υπάρχουν ε, άλλες ε, περιοχές που είναι πλέον κατάλληλες. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και βλέπω ότι η Επιτροπή Αναφορών ε, έχει μια τεράστια ευθύνη και υποχρέωση, αν κρίνω όπως είπατε. Κοιτάξτε, τα μέσα και οι τρόποι μας ε, είναι περιορισμένοι. Θα αφήσουμε φυσικά ανοιχτή την αναφορά. Αυτό είναι σαφές. Και νομίζω ότι εκ μέρους της Επιτροπής μας θα γράψω μια επιστολή στο Γάλλο Υπουργό Γεωργίας και... Μάλλον, συγγνώμη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος διόρθωση και... Θα αναφέρω τη συζήτησή μας στον Υπουργό, γιατί δεν ακούστηκε ούτε μία φωνή που να υπεστηρίζει το έργο αυτό, αυτή την επένδυση. Έτσι λοιπόν θα καταγράψω όλες αυτές τις απόψεις και θα ζητήσω εκ μέρους ε, της ε, Επιτροπής μας αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβει μία σαφή θέση και θα παρουσιάσω τις προσδοκίες ε, και της τοπικής κοινότητας, των κατοίκων αλλά και των πολιτικών. Θα τονίσω Επίσης ότι δεν ε, υπάρχουν ε, λόγοι ούτε κοινωνικοί, ούτε οικονομικοί, ούτε περιβαλλοντικοί για να συνεχιστεί αυτό το έργο. Φυσικά παραμένει ανοιχτή η αναφορά και θα επανέλθουμε αν χρειαστεί. Και κατανοώ ότι συμφωνείτε επί της διαδικασίας. Βλέπω ότι γνάφεται καταφατικά. Δεν διαμαρτύρεται κανείς. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και πολύ όλους όσους ήλθαν εδώ για να μας παρουσιάσουν την υπόθεση αυτή. Ας περάσουμε τώρα στο σημείο 19, αναφορά 13 κάθετος 2008. Έχετε το λόγο, κύριε πρόσωπε, των αναφερόντων, αλλά σας παρακαλώ μην μακρηγορήσετε άνω των 5 με 7 λεπτών. Monsieur le euh. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας κάνω εδώ την παρουσίασή μου. Η εταιρεία του ΙΦΑ του Σάνων Μα είπε ψέματα όταν κατέθεσε το αίτημά της, την αίτησή τη και έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρροή του υγροποιημένου αερίου. Θα σας δείξω ένα βίντεο δίλεπτο ενός ατυχήματος που έγινε το 87 στην έρημο της Νεβάδας και που δεν το έχουν δει πολλοί. Το ατύχημα έγινε από μια μικρή διαρροή 50 κυβικών μέτρων ύφα ενώ τα πλοία που το μεταφέρουν περιέχουν 5.300 φορές περισσότερο ύφα από το ποσότητα αυτή. Ο επενδυτής είχε δηλώσει ότι ως μέτρο προστασίας μπορεί κανείς να φύγει τρέχοντας, να κρυφτεί πίσω από δέντρα ή να κρατήσει μια εφημερίδα μπροστά στο πρόσωπό του. Αλλά ο Δόκτωρ Χέιβενς, που είναι ειδικό στο ΙΦΑ, είπε ότι ένα τέτοιο ατύχημα μπορεί να βλάψει ανθρώπους σε απόσταση τριών μιλίων από το πλοίο. Προς τα σχόλια της Επιτροπής για την αναφορά αυτή του Οκτωβρίου 2008 απαντούμε ως εξής. Για την, ε, για τον τεμαχισμό του σχεδίου, αν Board πλέον άλλα της Ιρλανδίας έχει ήδη δηλώσει ότι θα είναι, θα η αποτίμηση από την ε, υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν συμφωνούν οι δύο σχετικές αρχές μεταξύ τους για τις επιπτώσεις. Για την EIA δεν υπάρχουν όλες οι πληροφορίες στην μελέτη αποτίμησης, καθώς και αποτίμηση του κινδύνου στη θάλασσα από διαρροή ύφα. Ούτε σχέδιο άμεσης ανάγκης, γιατί στο σχετικό κυβερνητικό έγγραφο για τους κινδύνους του ύφα δεν δόθηκε δημοσιότητα. Και η υγροποίηση πάνω στο πλοίο και η ζημιά που θα αντιπροσώπευε μία διαρροή για τα δελφίνια δεν έχει αναφερθεί καθόλου. Για την στρατηγική περιβαλλοντολογική αποτίμηση πάνω από 10.000 άνθρωποι αφορούνται από το σχέδιο αυτό λόγω του κινδύνου που αντιπροσωπεύει η κίνηση των τάνκερ ΙΦΑ στην περιοχή εκείνη. Η δημιουργία λοιπόν του σχεδίου αυτού στο Δέλτα του Σάνων έχει σαν στόχο να εξάγει, να εξαγάγει το αέριο. Για τις τοποθεσίες τύπου Σεβέζο. Ο ελιμενισμός των πλοίων εκεί γίνεται με μεγάλο κίνδυνο γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί τα προβλεπόμενα από τη λεγόμενη οδηγία Σεβέζο και επιπρόσθετα θέλουμε αυστηρή εφαρμογή της προστασίας για αυτήν την πολύ ωραία ειδική διατηρητέα περιοχή. Γιατί υπάρχουν εναλλακτικές τοποθεσίες για την εγκατάσταση του κέντρου αυτού υγροποίησης. Μία από αυτές είναι η τοποθεσία της εταιρείας HERG για το υγροποιημένο αέριο κοντά στο Δουβλίνο. Εκτός από όλα αυτά μάθαμε ότι η εταιρεία Χέσ Άνων Ήφα είχε πληρώσει σχεδόν 500.000 ευρώ στην κυβερνητική εταιρεία Shannon Development πριν καν γίνει η μελέτη για την τοποθέτηση του κέντρου αυτού εκεί. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε θεωρούμε ότι η Ιρλανδική κυβέρνηση δεν είναι πια αντικειμενική στο θέμα αυτό και γι' αυτό ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ερευνήσει το θέμα σε μεγαλύτερο βάθος για να δούμε, για να γίνει για να δείτε αν είναι ακριβή αυτά που σας έχουμε υποβάλει και για να υπάρξει μια πιο συστηματική παρακολούθηση και επιτήρηση των πραγμάτων εκεί. Μια πρόσφατη ενωσιακή μελέτη για τη Γενική Διεύθυνση Τρέν κατέληξε ότι το αέριο είναι τμήμα του προβλήματος για την ε, θέρμανση του πλανήτη και όχι της λύσης. Στην Ιρλανδία Όποτε γίνεται αποτίμηση επικίνδυνων τόπων και τοποθεσιών, προσβλέπουν στα δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν κάνουν ειδική μελέτη για την Ιρλανδία. Και θεωρούμε ότι το κακό προηγούμενο που τέθηκε στο Milford Haven στο Ηνωμένο Βασίλειο θα επαναληφθεί και στην Ιρλανδία. Απλώς και μόνο γιατί είναι προηγούμενο. Ενώ δεν πρέπει να είναι προηγούμενο ο κακός σχεδιασμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα ο κύριος Ντεβέρτ, εκπρόσωπος της Κομισιόν. και τον αναφέροντα για τις πληροφορίες που μας χορήγησε σήμερα. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, τίθενται ορισμένα ερωτήματα, ιδιαίτερα ως προς την εφαρμογή των προβλεπωμένων για τις μελέτες αξιολόγηση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων όποτε σχεδιάζονται τέτοιες εγκαταστάσεις. Μερικά από αυτά τα προβλήματα είναι κοινά με των προηγουμένων αναφορών. Στην περίπτωση όμως αυτή σημειώνουμε ότι η άδεια δόθηκε το Μάρτιο 2008 ενώ στις προηγούμενες περιπτώσεις είχε ήδη αρχίσει η εφαρμογή. Έχουμε πρόσθετες πληροφορίες από τον αναφέροντα που ακόμη τις αποτιμούμε για να δούμε σε ποιο βαθμό έχει υπάρξει παραβίαση ή όχι της ενωσιακής νομοθεσίας. Και αν έχει υπάρξει θα θέξουμε το θέμα στις Ιρλανδικές Αρχές και θα πληροφορήσουμε και την Επιτροπή Αναφορών. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο Μπράιαν Κόλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον αναφέροντα που ήρθε ως εδώ για να κάνει την παρουσίασή του. Καταλαβαίνω ότι το θέμα αυτό αποτελεί πηγή προβληματισμού. Επίσης καλωσορίζω και τον, τους εκπροσώπους της αναπτυξιακής εταιρείας. Υπάρχουν όντως προβληματικά σημεία, όπως το αναφέρει και ο αναφέροντας, ο αλλά έγιναν όλα με τον προβλεπόμενο τρόπο. Προηγήθηκε διαδικασία διαβούλευσης και έναν μια ανεξάρτητη αρχή για θέματα χωροταξίας επίσης ε, γνωμοδότησε θετικά και το, το Συμβούλιο Χωροταξίας της περιοχής ήταν επίσης υπέρ. Έγινε προσφυγή στο ανώτατο δικαστήριο, η οποία όμως απορρίφθηκε. Το, απεφάνθη δηλαδή το δικαστήριο ότι η αρχή χωροταξίας είχε λάβει τη σωστή απόφαση. Οπότε τα θέματα που αφορούν ε, την, ε, την οδηγία σε Βεζό, την EIA ε, και την IPPC δεν έχουν βάση. Νομίζω ότι τίθεται θέμα παραπληροφόρησης. Μεγάλο μέρος του τοπικού πληθυσμού υποστηρίζει αυτή την, ε, την, αυτό το έργο, γιατί πρόκειται για στρατηγική επιλογή όσον αφορά τη διαφοροποίηση της, ε, του εφοδιασμού με κάψιμα και επίσης προάγει την κοινωνική, την κοινωνική ανάπτυξη σε αυτή την περιοχή της Ιρλανδίας. Θα το φυσικό αυτό αέριο θα ικανοποιήσει τις τοπικές ανάγκες και μπορεί ενδεχομένω και να εξαχθεί. Νομίζω ότι το θέμα της, της ευρύτερης διαβούλευσης είναι θεμητό όταν, όταν μιλούμε για διαβούλευση, στα 14 χρόνια της εμπειρίας μου στην ε, πολιτική ζωή της Ιρλανδίας, δεν έχω δει άλλο θέμα που να υποβλήθηκε σε τόσο ενδελεχή έλεγχο, διαβούλευση και συμμετοχή. Τέθηκαν διάφορα ζητήματα, όποτε τέθηκαν ερωτήματα δόθηκαν σαφείς απαντήσεις. Δεν υπήρξε κάποια παράτυπη απόκρυψη δεδομένων από την κυβέρνηση. Υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να κρίνει ότι, κάποια θέματα πρέπει, ότι πρέπει να διατηρηθεί μυστικότητα για κάποια θέματα. Αυτό είναι δεδομένο. Και ειδικά στην Ιρλανδία υπάρχει ειδικό κανονισμός που ενσωματώνει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να δημιουργηθεί προηγούμενο σε τέτοια θέματα. Δεν, οποιαδήποτε εξέλιξη στην Αγγλία ή σε άλλη χώρα δεν ε, προδικάζει την εξέλιξη στην Ιρλανδία ενός ανάλογου θέματος. Εδώ και αρκετά χρόνια είναι υποσυζήτηση αυτό το θέμα. Έχει χρησιμοποιηθεί κάθε δυνατότητα ε, αναστολής το, της εξέλιξης. Αυτή η διαδικασία που έχουμε, με την οποία ασχολούμαστε τώρα, της υποβολής αναφοράς στην Επιτροπή Αναφορών, είναι ακόμα μια, ε, συνιστά ακόμα μια καθυστέρηση. Ευχαριστώ. Η ερώτησή μου είναι αν θέλει κάποιος να λάβει το λόγο. Ίσως πρέπει να θέσουμε πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις στην Επιτροπή. Να ζητήσουμε ίσως διευκρινήσεις. Ο κύριος σας δίνω το λόγο να απαντήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα σχόλια του Ξιότιμου μέλου σχετικά με αυτή την αναφορά έχουν κάποια βάση, έχουν βάση. Δεν μπορώ να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα δεδομένα που μου κοινοποίησε ο αναφέρον. Σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να κάνω κάποιο περαιτέρω σχόλιο. από, από την άποψη των βουλευτών ακούσαμε τον κύριο Κρόλι, Ήταν πολύτιμες οι, θέσεις, οι απόψεις σας. Αν θέλει κάποιος άλλος το λόγο, ίσως ξανά εσείς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε μια, μια παρεμφερή αναφορά με τις δύο προηγούμενες δεδομένου ότι υποστήριξα στεναρά τις δύο προηγούμενες, δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω και αυτήν. Δεν είναι της αρμοδιότητάς μου το θέμα, δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες, αλλά νομίζω ότι τα δεδομένα που μας έχουν παρασχεθεί είναι υπεραρκετά. Και πιστεύω επίσης ότι ίσως πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά μέχρι να αποφανθεί και η Κομισιόν. Ε, πρόεδρε, δεδομένων όλων όσων ακούσαμε εδώ, θα ήθελα η Επιτροπή, αντί να περιμένει για την επόμενη συνεδρίαση, να σας ενημερώσει σχετικά με την απάντηση που θα δώσει ως προς τα συμπληρωματικά στοιχεία που επέβαλε ο, επέβαλε ο αναφέρον στην κυρία Εύανς και τον κύριο Κόουλ, Κρόουλ. Είτε θα παραμείνει ανοιχτή, είτε θα περατωθεί η εξέτασή της. Οπότε αντί να περιμένουμε για την επόμενη συνεδρίαση, νομίζω ότι θα είναι πιο παραγωγικό αν καταλήξουμε τώρα. Υπήρχαν, υπήρξαν διαφορές μεταξύ των όσων είπε η κυρία Evans και ο κύριος Κρόλι. Οπότε η καλύτερη λύση είναι μπορούμε αφενός να, αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να περιμένουμε τις απαντήσεις της Επιτροπής. Κύριε Κρόουλη, εσείς ε, συμφωνείτε με αυτό, να παραμείνει ανοιχτή δηλαδή η αναφορά μέχρι να μας δώσει την απάντηση η Επιτροπή. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος να παραμείνει ανοιχτή. Αν μπορεί η Επιτροπή να δώσει τώρα την απάντησή της στην Επιτροπή Αναφορών, θα ήταν καλύτερο αν μπορούν τη, τώρα εδώ να δώσουν την απάντηση, καλό θα ήταν να περατωθεί επιτέλους η εξέταση αυτής της αναφοράς, γιατί έχει τραβήξει ήδη σε μάκρο αρκετά και δεν είναι δίκαιο ούτε για τους εμπλεκομένους, τους κατοίκους της περιοχής. Νομίζω ότι ε, προσωπικά είμαι αντίθετος στην διατήρηση αυτής της αναφοράς. Οι προβληματισμοί του κυρίου Κρόλη πρέπει προφανώς να ληφθούν υπόψη. Η συνήθις διαδικασία είναι η εξή. Αν η Επιτροπή Κομισιόν είναι της άποψης ότι θέλει να πει κάτι ακόμα σχετικά με κάποιο θέμα, σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, εμείς περιμένουμε. Αλλά προφανώς πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο παράγοντας χρόνος. Ίσως μπορούμε λοιπόν να ζητήσουμε από την Κομισιόν να αποστείλει τις απαντήσεις της σε εμάς, στις ερωτήσεις που τέθηκαν σήμερα. Πριν από τη λήξη της θητείας του τρέχοντος κοινοβουλίου και έτσι ώστε να περατωθεί τελικά και η εξέταση της, της αναφοράς. Η Κομισιόν ε, άφησε να εννοηθεί ότι θα ήθελε να συμπληρώσει κάτι Κοιτάξτε, μας έχουν μείνει έξι εβδομάδες ακόμα για τη θητεία και με κάθε σεβασμό απέναντι στην Κομισιόν, ε, εγώ ξέρω ότι συνήθως ε, χρειαζόμαστε πάνω από τέσσερις εβδομάδες συνήθως για να έχουμε καμία απάντηση και δεν ξέρω αν θα έχουμε χρόνο για να κλείσουμε αυτή την αναφορά. Και πάλι εσεί ω πρόεδρο πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη σοφία σα ε, για να δούμε πώ θα καταλήξουμε. Αλλά νομίζω ότι δεν θα ήταν σωστό να μην ήταν η Κομισιόν σε θέση να μας δώσει απαντήσεις, ενώ εκ των προτέρων γνώριζε τι θα συζητούσαμε εδώ σε αυτή τη συνεδρίαση. Αν ε, μπορώ να πάρω το λόγο, Πρόεδρε, εκ μέρου σα, Ο κανόνας ε, είναι να ήταν να διατηρούμε ανοιχτή ε, την αναφορά προκειμένου να λαμβάνουμε απάντηση. Μάλλον αυτό είναι το προηγούμενο και νομίζω ότι ο πρόεδρος δεσμεύεται, αλλά μάλλον ε, μπορούμε να έχουμε σύντομα μια επίλυση του ζητήματο. Βλέπω η Κομισιόν γνέφει καταφατικά, επομένως ε, θέλουμε να επιταχύνουμε τι απαντήσει και να μπορέσουμε να συζητήσουμε εκ νέου με του αναφέροντες και να λάβουμε κάποια απόφαση. Πρέπει λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή έτσι, αυτή, συγγνώμη αναφορά αυτή και τώρα... Σας δω συγγνώμη πρόεδρε που πήρα το λόγο, αλλά καταλαβαίνετε ήταν πολύ σαφής ε, η λόγη. Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά μήπως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα σε δύο εβδομάδες θα μπορούσε να μας στείλει την απάντηση, θα ήταν δυνατό κάτι τέτοιο. Uh, so, yeah. Θα προσπαθήσουμε. Επειδή υπάρχουν ε, πάρα πολλά τεχνικά στοιχεία, χρειάζεται να γίνει περαιτέρω τεχνική αξιολόγηση των πληροφοριών, αλλά θα σας... Ε, θα προσπαθήσουμε να σας τη στείλουμε. Εντάξει, ας ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς ε, προσπαθούμε να αποφύγουμε την ψηφοφορία, αλλά αν τα μέλη της Επιτροπής ε, απευθύνουν έκκληση εδώ να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά, συνήθως αυτό κάνουμε χωρίς να υπάρχει μια ψηφοφορία. Γιατί η ψηφοφορία είναι η τελική μας λύση και σπανίως προσφεύγουμε σε αυτήν. Πάμε τώρα στην επόμενη αναφορά, 74 του 2008. Είναι μαζί μας και ο αναφέρον. Η αναφέρον μάλλον, η αναφέρουσα Μαρία Χεσούς Πέρεξα Κορέτα, αλλά και ο κύριος Αμάλιο Δεμαριτσαλάρ. Δέκα λεπτά έχετε μαζί, από κοινού. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλό σας απόγευμα. Συγγνώμη. Καλησπέρα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφορών που έκανε παραδεκτή την αναφορά και δέχτηκε να εξετάσει αυτή την αναφορά για την προστασία του πολιτιστικού ε, και περιβαλλοντικού βάλλοντος. Ε, ε, τοποθεσία της Νουμάνσια κατά 1130 μέτρα, βρίσκεται σε 1130 μέτρα υψόμετρο, 8 χιλιόμετρα από την πόλη της ε, Σόρια. Ε, ο θύλακας αυτός περικυκλώνεται από μικρές ιστορικές τοποθεσίες όπου Σκυπίωνα σε ίδρυσε τους κατοβλισμούς τα έτη 134 133 π.Χ. και ε, αυτή η τοποθεσία στην ε, λατινική αλλά και παγκόσμια λογοτεχνία ε, αποτέλεσε το σύμβολο της αντίστασης και ενός λαού, ενός λαού που υπεράσπισε την ελευθερία του αν ε, σήμερα και από την τοποθεσία αυτή μπορεί ο επισκέπτης να δει ολόκληρο το τοπίο που ήδη οι Βεροκέλτες από το 154 π.Χ. όταν ξεκίνησαν ε, τους κελτεβερικούς πολέμους μέχρι την ολική καταστροφή το 133 π.Χ. μπορούσαν ε, να δουν ε, όλο αυτό το τοπίο, τότε τα σχέδια ε, των Δήμων Γκαρά Ισόρια σημαίνει ότι θα έχουμε αναπόδραστη καταστροφή του τοπίου του ποταμού του Έρου. Σκοπεύεται ουσιαστικά να υπάρχει κατασκευή ενός συνόλου κατοικιών που θα περικυκλώνουν τον ρωμαϊκό καταφλισμό του Άρτο Ρεάλ ε, και ε, Επίσης θα κατασκευαστεί ένα βιομηχανικό σύμπλεγμα, Σόρια 2, ε, που το βλέπετε με το ροζ και θα βρίσκεται μεταξύ της Ρουμάνσια και του Ρωμαϊκού κύκλου του Σκυπίωνα, ενώ σε 400 μέτρα βρίσκεται ο Ρωμαϊκός καταφυλισμός της Ράσα. Βλέπετε εκεί το βιομηχανικό σύμπλεγμα 2 εκεί έχουμε την πόλη Σόρια, και βλέπετε και τις ε, κατοικίες του Γκαράη. Εδώ βρίσκεται η Νουμάνσια και στη συνέχεια η κίτρινη γραμμή δείχνει που είναι ο τείχος που διάταξε ο Σκυπίωνος να κατασκευαστεί ε, προκειμένου να προστατεύσει ε, την πόλη μάλλον συγγνώμη, να πνίξει την πόλη, να την πολιορκήσει και να μην φτάνουν οι προμήθειες. Έτσι λοιπόν ε, βρισκόμαστε στα 400 μέτρα από τον ε, καταβλισμό της Ράσα και την, ε, την Ρωμαϊκή Εκκλησία και το καμπαναριό του Σαν Χουάν και αυτά έχουν διακηρυχθεί η πολιτιστική, παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Επίσης ε, υπάρχει και ένα νεκροταφείο ε, στη ζώνη αυτή ε, και στη ζώνη αυτή υποτίθεται ότι έχουμε μεγάλη κελτική παράδοση. Επομένως βλέπετε ότι θίγεται ένας τόπος όπου έχουμε μεγάλη ιστορική και λογοτεχνική παράδοση και ε, γι' αυτό αυτό το τοπίο που έχει μείνει ε, σχεδόν αναλύωτο για 2.000 χρόνια συνεννοών στον 21ο αιώνα τελικά θα καταστραφεί από τον άνθρωπο ενώ τον 21ο αιώνα έχουν γίνει τόσες μεγάλοστομες περιβαλλοντικές ε, δηλώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και, έχει, και έχουμε εγκρίνει και σημαντική νομοθετική και έχουμε κάνει σημαντικό νομοθετικό έργο για την προστασία της πανίδας και της φλωρίας. Είναι παράδοξο λοιπόν ακριβώς γύρω από την Ουμάνσια ναι, και τη Σόρια, μια περιοχή όπου υπάρχουν τόσο μεγάλες ε, ε, παιδιάδες και ενώ υπάρχουν άλλες περιοχές που μπορούν να αναπτυχθούν τέτοια έργα, Ακριβώ ε, παρουσιάζεται αδικαιολόγητα αυτό το έργο. Τι νόημα έχει λοιπόν να κατασκευαστούν 780 κατοικίες και 300 ξενοδοχειακές και μονάδες ξενοδοχειακές. μέσα σε ένα ε, στο στο Σότα Ντεγκαράι, όπου έχουμε μεγάλο φυσικό πλούτο με πάρα πολλά είδη δέντρων και υπάρχουν και διάφορα είδη πτηνών που φωλιάζουν εκεί. Ε, και η κατασκευή 288 κατοικιών επίσης στο Γκαράι, γύρω από το ρωμαϊκό κατευνισμό. Παρακαλώ δείτε την επόμενη διαφάνεια. Εδώ ε, μιλάμε ε, για μία κατασκευή που δεν έχει ακόμη αρχίσει ε, την κατασκευή γιατί υπάρχει προσφυγή από ε, βουλευτές ε, του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Ισπανίας. Επίσης, βλέπετε εδώ ένα άσπρο σημείο ε, και εκεί άρχισαν οι ανασκαφές στις αρχές ε, του 20ου αιώνα και εκεί έχει γίνει ένα είδος εικονικού καταφυλισμού και βλέπετε ε, σαν να ήταν εκεί το μέρος όπου υπήρχαν οι λεγεώνες Όμως εδώ τώρα ε, ήθελαν εδώ να κάνουν αποκατάσταση ε, του, ε, του αρχαιολογικού χώρου και ακολουθήθηκε μία εντελώς παράνομη διαδικασία. Ε, εδώ στο Άλτο Ρεάλ δεν έγιναν σκαφές, αλλά έχουν αρχίσει να γίνονται εγκαταστάσεις όπως τις τηλεφώνικα λόγου χάρη. γνωρίζουμε ότι αυτές οι κατασκευές των χιλίων κατοικιών εδώ έχουμε και πάλι το Alto Real και στο βάθος ε, το Σέρο Δελαμουέλα, όπου έχουμε την πόλη της Νουμάνσια. Η κατασκευή λοιπόν αυτών των κατοικιών ε, δίπλα σε μια μεσαιωνική πόλη αλλά και ε, κτηρίων ε, θεσμικών ε, σημαίνει ότι θα υπάρχει πολύ σοβαρή υποβάθμιση, υποβάθμιση η οποία θίγει ένα ιδιαίτερο περιβάλλον από κάθε σκοπιά και τώρα κατασκευαστεί αυτό το σώριο εντό αυτό το βιομηχανικό σύμπλεγμα σε μια τοποθεσία πιο υπερυψωμένη ουσιαστικά είναι παράλογο ε, γιατί υπάρχει, ε, υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι ε, τριγύρω που θα μπορούσε να κατασκευαστεί ένα τέτοιο σύμπλεγμα και μάλιστα ήδη κατασκευάζεται ένα άλλο τέτοιο βιομηχανικό σύμπλεγμα εκεί κοντά που λέγεται Μπαλκόρια ο αντίκτυπος που θα έχει αυτό το έργο ουσιαστικά καταργεί από τις μελλοντικέ γενιές ε, το να απολαύσουν ε, μια τέτοια πολύ σημαντική αρχαιολογική τοποθεσία. Έχουν ε, παρουσιαστεί άλλες εναλλακτικές λύσεις που ε, μπορούν να συμβάλλουν ε, στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής με την ταυτόχρονη προστασία της πολιτικής της κοινωνιάς. Έτσι λοιπόν απευθύνουμε έκκληση στη Ισπανική κυβέρνηση, στη Χούντα Δικαστήγερεών ε, και στο Ισπανικό Υπουργείο Πολιτισμού να λάβουν υπόψη όλα τα επιχειρήματα και τις αποδείξεις που έχουμε αναφέρει τις γνωμοδοτήσεις από διάφορα ε, από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, το Νίκο του Βελάσκες και διάφορους άλλους οργανισμούς. Έχουμε επίσης συλλέξει πάνω από 12.000 υπογραφές για να οθήσουμε τις αρμόδιες αρχές στο να ζητήσουν να κηρυχθεί η τοποθεσία της Νουμάντσια ως περιοχή πολιτιστικής κληρονομιάς, παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Εμείς ε, θέλουμε να ε, ευαισθητοποιήσουμε τους υπευθύνου, τους ηθήνοντες, να σκεφτούν ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης που να μην θέτει σε κίνδυνο την κληρονομιά μας. Πολύ γρήγορα για να δείτε τις επόμενες φωτογραφίες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα, επόμενο, ομιλητής, ε, κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, εδώ εκπροσωπώ την οικογένειά μου, αλλά και τον εαυτό μου και σα ευχαριστώ για την ακρόαση αυτή. Θέλω να καταγγείλω την ε, κατασκευή αυτού του βιομηχανικού συμπλεγματο ΣΟΡΕ 2 ε, στη δική μα γη και αυτό έχει καταγγελθεί από διάφορα Ινστιτούτα και Ιδρύματα παγκόσμιου Βεληνικού. Πιστεύω ότι τον 21ο αιώνα η δημοκρατία δεν μπορεί μπορεί να επιτρέψει να γίνει αυτή η κατασκευή σε μια τοποθεσία όπου έχουμε 7 7 ε, ε, αρχαιολογικές ε, τοποθεσίες. Πριν λίγο καιρό ελήφθησαν κάποια αντισταθμητικά μέτρα για την υπεράσπιση του αρχαιολογικού χώρου της Νομάνσια. Ο κύριος Χάμερστάιν μάλιστα πριν λίγο καιρό ανέφερε, έκανε μια καταγγελία βάση της μιας οδηγίας προστασίας του περιβάλλοντος γιατί θεώρησε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να προάγουμε τον τουρισμό. Μάλιστα, η διγεια 2001 2001-42 πρέπει να αναφερθεί από μένα, γιατί ουσιαστικά αναφέρεται στην επίπτωση που έχουν ορισμένα σχέδια και έργα στο περιβάλλον. Επίσης, ε, πριν ε, να υιοθετηθούν πλήρως τα προγράμματα των ε, κρατών μελών, θα πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση για τη χρήση του εδάφους. Βασικά, το έγγραφο του Δήμου είπε ότι θίγεται ένας πάρα πολύ μικρός χώρος. Συγγνώμη, πρέπει να διαβάσετε πιο αργά για τη διερμηνία. Λέει στο έγγραφο αυτό ότι καθώς η Σόρια βρίσκεται πάρα πολύ κοντά και καθώς ε, διαιρείται η ζωνή. Λυπάμαι. Λοιπόν, έλεγα ότι λέει το έγγραφο ότι από την Ουμάνσια βλέπουμε το κάστρο ε, και το Μόρτι Δελασάνη μας. Πάντως ο Δήμος είναι εντελώς ε, αντίθετος στη 2001-42 για τους εξής λόγους δεν έχει ε, εξεταστεί η περιβαλλοντική διαδικασία που απαιτεί οδηγία για την εκπόνηση και την οριστική έγκριση του ε, αντικτύπου του σχεδίου, συγγνώμη, επίσης δεν έχει υποβληθεί η περιβαλλοντική έκθεση προβλέπεται στην ε, οδηγία Τρίτο, η περιβαλλοντική διαδικασία της οδηγίας τουλάχιστον ήταν υποχρεωτική, καθώς το σύμπλεγμα φύγει μια πολύ σημαντική ποσότητα του εδάφους, 116 εκτάρια. Η οδηγία υποχρεώνει στο να γίνει η προηγούμενη περιβαλλοντική διαδικασία έγκριση των σχεδίων που επιτρέπουν ε, την δημιουργία μελλοντικών σχεδίων, όπως είναι το Σόρια 2.4. Μιλάμε για μια έκταση 116 εκταρίων, ε, όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει εκεί αυτή, αυτό το έργο και ε, πραγματικά οι Ισπανικές αρχές δεν έχουν παρουσιάσει κανένα λόγο γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι το 5. Ε, θα μπορούσαμε να έχουμε τη μηδενική εναλλακτική και αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να μην κατασκευαστεί ε, αυτό το σύμπλεγμα γιατί ε, θα θίξει ανεπανόρθωτα την περιοχή μέχρι σήμερα. Ε, το Ισπανικό κράτος δεν έχει κάνει τίποτα για να υπερασπίσει την εφαρμογή του νόμου 1-2006-28 Απριλίου, ε, ούτε έχει μεταφέρει την οδηγία 2001-42 στο εσωτερικό του δίκαιο. Επίσης, το ανώτατο δικαστήριο της ε, Καστίγια Λεόν ε, έχει προβεί σε δικαστική απόφαση παρόμοια περίπτωση 29 Σεπτεμβρίου 2006 με ε, παρόμοια επιχειρήματα γιατί είχε πει ότι έπρεπε να γίνει νέα αναθεώρηση του σχεδιασμού. Δεύτερον, ότι πρέπει να γίνει πρώτα, να είναι γνωστός ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος, προκύπτει από την ταξινόμηση της χωροταξίας που προβλέπει βλέπετε στο σχέδιο. Επίσης, σε ε, συγκεκριμένη περίπτωση όταν ε, ε, τέτοια έργα θίγουν έκταση άνω των 100 εκτερίων είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ταξινόμηση του εδάφους ως περιορισμένο έδαφος όπου μπορεί να χτιστεί. Επίσης, να σας ε, αναφέρω ότι κοντά στη Σόρια υπάρχουν και άλλες ιστορικές νομοθεσίες και πραγματικά εμένα ε, με εκπλήσει ότι οι Ισπανικές αρχές ε, απέναντι σε αυτό το θέμα πραγματικά σιωπούν. Η Νουμάνσια είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο και επίσης να σας πω ότι υπάρχει κατάχρηση εξουσίας και θεσμική κερδοσκοπία. Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά έτσι είναι. Και αυτό το θέμα μας ε, θίγει εμάς και ως πολίτες, θίγει την οικογένειά μου και δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε μπροστά στις τεράστια εξουσία των θεσμών. Πραγματικά εδώ ε, και τα δικά μας συμφέροντα υπερασπιζόμαστε, τα νόμιμα συμφέροντα αλλά και τα συμφέροντα όλων των πολιτών και στην Ισπανία αλλά και παγκοσμίως και γι' αυτό θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε ε, να δούμε ένα βίντεο 1,5 λεπτού για να κλείσουμε αυτή την ε, παρουσίαση. Να σας πω ότι αγωνιζόμαστε έτσι ώστε ε, νομικά να επιστρέψουμε στο να κατηγοριοποιηθεί αυτή η περιοχή ως μια περιοχή αγροτική γιατί τώρα έχει λάβει το χαρακτηρισμό της βιομηχανικής. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Empieza con unas buenas... Λοιπόν, βλέπετε εδώ κάποιες ε, τελικά βλέπετε κάποια φαγητά, κάποιες σπεσιαλιτέ. Segundo, para los golosos una tentación difícil de resistir.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 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Κομισιόν μπορεί απλώς να εξετάσει το θέμα λαμβάνοντας υπόψη την κοινωτική νομοθεσία στο περιβαλλοντικό τομέα. Η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Περιβάλλοντος είναι η αρμόδια για τη διαβούλευση σε ό,τι αφορά τώρα το περιφερειακό πρόγραμμα ε, της ε, ε, πόλης της Μεσαιωνικής ε, να σας πω ότι αυτό το project έχει ήδη μελετηθεί στα πλαίσια της 2007-2021-25 2025 αναφορας και η Κομισιόν δεν μπόρεσε να εξεύρει ότι υπάρχει παραβίαση της ε, περιβαλλοντικής κοινωτικής νομοθεσίας. Τώρα για το ΣΟΡΙΑ 2. λόγω κοινοβουλευτική ερώτηση, αλλά και λόγω των νέων καταγγελιών που λάβαμε σχετικά και λόγω των αναφορών, η Κομισιόν ξεκίνησε μια διαδικασία έρευνας για το θέμα αυτό και το αποτέλεσμα των πληροφοριών που λάβαμε από τις Ισπανικές Αρχές μας οδήγησε, ήταν το εξής, μας οδήγησε σε κάποια συμπεράσματα σε σχέση με το αν παραβιάζεται η οδηγία για τους οικοτόπους να σας πω ότι το σχέδιο καθώς ε, βρίσκεται στα βορειοανατολική ισορία, ε, δεν θίγει κάποιους ε, προστατευμένες, κάποιες προστατευμένες περιοχές, ούτε κάποιους τόπους που έχουν χαρακτηριστεί κοινοτικού ενδιαφέροντος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη 2001-42 οδηγία για την αξιολόγηση του αντικτύπου ορισμένων σχεδίων στο περιβάλλον, η οδηγία αυτή προβλέπει στο άρθρο 3, παράγραφος 3, ότι τα προγράμματα και τα σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 που έχουν να κάνουν με την χρήση μικρών περιοχών σε τοπικό επίπεδο και την μικρή τροποποίηση σε σχέδια που αναφέρονται έχουν περιβαλλοντικό αντίκτυπο μόνο αν αποφασίσουν τα κράτη-μέλη ότι έχουν τέτοιο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σημαντικό. Οι Ισπανικές αρχές ε, είπαν ότι δεν χρειάζεται να γίνει μελέτη αντικτύπου και αυτό έχει δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Καστίγια Ελαιών ε, στο τεύχος 81 και είπαν ε, ότι τα εκτάρια αυτά έχουν ε, ε, θεωρηθεί ως μια αγροτική περιοχή η τροποποίηση θα σήμαινε ότι μόνο το 0,1% αυτής της γης που έχει χαρακτηριστεί ως αγροτική περιοχή θα θυγόταν και θα είχαμε αύξηση 26% μόνο του βιομηχανικού εδάφους. Επίσης να επισημάνουμε ότι η αιτιολογημένη απόφαση επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν καταλογοποιημένοι αρχαιολογικοί θύλακες υπό την φύλαξη των τη λογημένη απόφαση που ανέφερε προηγουμένω, αναφέρει ότι το μερικό σχέδιο του βιομηχανικού πλέγματο θα αξιολογηθεί από περιβαλλοντική σκοπιά σύμφωνα με το νόμο της 28 Απριλίου 2006 για τον αντίκτυπο των προγραμμάτων και των σχεδίων στο περιβάλλον. Αυτός ο νόμος μεταφέρει στο Ισπανικό Ιστορικό Δίκαιο τη 2001-42. Επίσης έχουμε την ε, οδηγία του 85 και δυνάμεις αυτής ή Κομισιόν ε, δεν μπόρεσαν να βρουν ότι υπάρχει παραβίαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Από την άλλη, η Κομισιόν έλαβε γνώση της εξέτασης μιας προσφυγής σε διοικητικό επίπεδο, αλλά και το ότι έχουν ληφθεί κάποια ασφαλιστικά μέτρα και για το λόγο αυτό θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να συνεχίσει την έρευνα που έχει ξεκινήσει γιατί επί της ουσίας ε, του ζητήματος δεν, έχουν υπάρξει δεν έχει υπάρξει λήψη αποφάσεων. Ευχαριστώ. Κύριε Δεμέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με δέχεστε εδώ στην Επιτροπή σας, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει και με απασχολεί. Καθώς και εγώ προέρχομαι από τη Λεόν και είμαι και Σπανός φυσικά, την στη Λεόν. Συγγνώμη, έχω κάποιους περιορισμούς ε, από σωματική σκοπιά. Θα ήθελα να χαιρετήσω την κυρία Πέρεξ και τον κύριο Μαριτσαλάρ τους συμπατριώτες μου και να πω ότι έχουμε σημεία στα οποία είμαστε σύμφωνοι αλλά και σημεία στα οποία διαφωνούμε. Οι αναφορές ε, τις οποίες ε, εξετάζουμε αναφέρονται σε δύο έργα τα οποία παρόλο που είναι εντελώς ανεξάρτητα τελικά εμπλέκονται στις ε, αναφορές και στις καταγγελίες που παρουσιάζονται σε αυτήν την Επιτροπή. Το ένα είναι το ε, η κατασκευή του συμπλέγματος Σόρια 2 και το άλλο είναι η Μεσαιωνική πόλη. Μεταξύ των δύο υπάρχει μια γεωγραφική απόσταση 90 χιλιόμετρων ή περισσότερων γιατί έχουμε και το ποτάμι όπως είδατε και πάνω από χιλιόμετρα αν μιλήσουμε για προγραμματικές θέσεις χρήσης ή εκμετάλλευσης η καταγγελία σε σχέση με την ε, περιβαλλοντική πόλη εξετάστηκε από την Κομισιόν δύο φορές όπως ακούσαμε το 2007 ε, και το 9, και η Κομισιόν θεώρησε ότι αυτό το έργο δεν παραβιάζει την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία ούτε την 9243 ε, ούτε την οδηγία 402 ουσιαστικά μιλάμε για την κατασκευή, μια, για μια θεματική κατασκευή όπου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αποτελούν θεμελιώδες συστατικά ενός ε, σχεδίου ε, αηφόρου ανάπτυξης για τη Σόρια και την ευρύτερη περιοχή. Επίσης, ε, η Χούντα της Καστίγια Λεών κήρυξε ότι αυτό το έργο παρουσιάζει ιδιαίτερο περιφερειακό ενδιαφέρον και δεν έχουν υπάρξει υπάρξει αποδείξεις ότι θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο δίκτυο Natura 2000. Και μάλιστα δηλώνεται ότι έχει ληφθεί υπόψη ο πιθανός αντίκτυπος στο νερό, στον αέρα, στο κλίμα, στο έδαφος, στο τοπίο, στην πανίδα, στη χλωρίδα, στα υλικά αγαθά και στην αρχαιολογική κληρονομιά και στη φύση. Ε, και σε ό,τι αφορά την καταγγελία που έχει να κάνει με το Δημοτικό Σύμπλημα Σόρια 2, εγκρίθηκε ε, από τα 20 από τα 21 εταιρικά μέλη του Δήμου της ε, Σόρια. Ένας απόσχε και οι 20 το ενέκριναν. Εγώ θα ήθελα να σας στήσω και θα ήθελα να παρακαλέσω να βάλετε στο φάκελο το διάταγμα 1625, αριθμός 201 της Καστήγια Ελαιών. Η Κομισιόν ζήτησε και απέκτησε επαρκείς πληροφορίες που τις επέτρεψαν να δώσει τις κατάλληλες πληροφορίες που μόλις ακούσαμε. Δεν υπάρχουν λοιπόν αρχαιολογικοί θύλακες που θίγονται και το μερικό σχέδιο θα υποβληθεί σε περιβαλλοντική αξιολόγηση. Υπογραμμίζω και το λέω για την Κομισιόν, δεν υπάρχει παραβίαση πελοβητικής νομοθεσίας περιβαλλοντικής κοινοτική νομοθεσία. Έτσι λοιπόν, Πρόεδρε, αυτό είναι μια άλλη διαφορετική σκοπιά από αυτή που ακούσαμε, μια άλλη άποψη. Φυσικά είναι σεβαστή η άποψη, αλλά νομίζω ότι τελικά πρέπει να δούμε και ποιο είναι το κριτήριο και η κρίση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χαμερστάιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλές φορές Μιλήσαμε για σημαντικές πολιτιστικές τοποθεσίες ε, που δεν λαμβάνονται υπόψη στην ε, περιβαλλοντική μελέτη που Αναφέρουμε την περίπτωση της ε, Τάρα. Εδώ μιλάμε για μια αρχαιολογική περιβάλλουσα τοποθεσία. Η αλήθεια είναι ναι, ότι το έργο αυτό δεν γίνεται επάνω στην τοποθεσία. Αυτό έλειπε άλλωστε. Αλλά πραγματικά έχει επιπτώσεις στο τοπίο το οποίο έχει τόσο πολύ μεγάλη αξία που εκατοντάδες εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη και οργανώσεις που την πιο σημαντική πολιτιστική κληρονομιά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούν να υπάρξει πρόληψη. Η οδηγία στρατηγικής αξιολόγησης θα έπρεπε ε, να αξιολογήσει αυτό τον αντίκτυπο στο τοπίο επιπρόσθετα η μορφή τη σύναψη τη σύμβαση. Εδώ δεν έχουμε κάποιον από την εσωτερική το σχολιάσει. Το πώ έγινε ε, η ανάθεση λοιπόν αυτών των δημοσίων έργων αυτό το ε, δημόσιο συμφέρον, όπως αναφέρθηκε. Πώς αιτιολογήθηκε, αιτιολογήθηκε σύμφωνα με τον νόμο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη Σύναψη Συνέσεων. Ε, εδώ μιλάμε ε, για την κατασκευή κατοικιών, οι οποίες διαφημίζονται επικαλούμενες στο ότι βρίσκονται κοντά σε αρχαιολογική περιοχή. Επίσης, αυτό θίγει και την το, το ποτάμι ε, ουσιαστικά του Ντουέρο και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου το περιβαλλοντικό δίκαιο ως προς την αξιολόγηση και ως προς τη σύναψη συμβάσεων και ως προς την χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ είναι δυνατόν οι αρχέ Καστιγελών να ανακοινώνουν ότι αυτό το έργο έχει χρηματοδότηση 30 δισεκατομμυρίων, να μου το σχολιάσει αυτό η Γενική Διεύθυνση περιφερειακή πολιτική ενώ δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση. Και λένε ότι έχει κοινοτική χρηματοδότηση όταν κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Βρισκόμαστε λοιπόν ενώ, ενώπιον μιας, ε, νομοθε, ενός νομοθετικού κενού. Και εσείς πρόεδρε πολύ καλά μπορείτε να το εκτιμώσετε αυτό. Εδώ μιλάμε για μια πάρα πολύ γνωστή τοποθεσία σε όλη την Ευρώπη. Εγώ πήγα εκεί, μετέβηνε εκεί και θα δούμε και βλέπουμε ότι αν κάποιος ε, γύρω γύρω βάλει όλα αυτά τα κτίρια τότε δεν θα είναι ίδια η αξία της ιστορικής τοποθεσίας. Αυτό είναι ηλίου φαϊνότερον. Ευχαριστώ κυρία Γκαρσία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 σε αυτή την Επιτροπή. Ε, ε, το σχέδιο ΣΟΡΕΑ 2 προωθείται από το Δήμο Καστίγια Ελαιών μέσω της Χεστουρκάλ και το Δημαρχείο της ΣΟΡΕΑ το 2005 έδωσε, ε, έθεσε στη διάθεση της Χεστουρκάλ που είναι η δημόσια επιχείρηση του Δήμου Καστίγια Ελαιών για την διαχείριση της χωροταξίας όταν ζητήθηκε βοήθεια δηλαδή ε, και η τεχνική της Καστίγια Λεών διάλεξαν την οριστική τοποθεσία. Η επιλογή της περιφερειακής κυβέρνησης ήταν ε, σαφής όπως ε, βλέπετε και στα έγγραφα της προηγούμενης θητείας των νοτικών Συμβουλίων δηλαδή είτε θα επιλεγόταν αυτή η τοποθεσία είτε καμία. Η θέση της σημερινής κυβέρνησης ήταν να αναπτυχθεί το δεύτερο στάδιο του συμπλέγματος της Βαλκούρβα, αλλά εφόσον λήφθηκε, από τότε που ελήφθηκε η απόφαση αυτή, ε, σήμερα τι γίνεται. Το Δημαρχείο της Σόρια, γνωρίζοντας ε, πως, ότι λείπει ε, ότι δεν υπάρχει έδαφος για κατασκευή βιομηχανικών συμπλεγμάτων δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτό το έργο. Πραγματικά αναγνωρίζει ότι ίσως να μην είναι η καλύτερη επιλογή ε, η επιλογή αυτού του συγκεκριμένη τοποθεσία, αλλά όχι για τους λόγους που αναφέρατε, δηλαδή πολιτιστικούς, ε, αρχαιολικούς, περιβαλλοντικούς κτλ, αλλά για λόγους πόρων ο Δήμος Καστίγια Λεών έχει θέσει κάποια θέματα που θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε. Η περιοχή όπου θα γίνει η κατασκευή είναι ε, μια περιοχή η οποία δεν προστατεύεται ούτε περιβαλλοντικά ούτε αρχαιολογικά. Τα ε, ρήπια της ε, Ρουμασία δεν βρίσκονται στο Δήμο της Όρια αλλά στον Καράι. Στις 4 Οκτωβρίου 2008 έγινε μια συνεδρία του Δημού και ε, ενημερώνει ότι ε, στο πλαίσιο ε, αυτής της τοποθεσίας όπου θα χτιστεί το Σόρια 2 δεν θίγεται καμία αρχαιολογική περιοχή. Ίσως υπάρχει κάποιος αντίκτυπος σε ό,τι αφορά το τοπίο αλλά παρουσιάζεται μία πρόταση να ε, φυτευτούν κάποια δέντρα, το χάρη, έτσι ώστε ε, να κρύβεται ένα μεγάλο μέρος ε, του συμπλέγματος που μπορεί να φαίνεται από μακριά. Επίσης, θέλω να δηλώσω εδώ ότι το Δημαρχείο της Ωρία βρίσκεται στην απόλυτη διάθεσή σας για να σας παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να ξεκαθαρίσει το ζήτημα αυτό. Ο Δήμος της Ωρία πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί το έργο αυτό, το βιομηχανικό σύμπλεγμα και εμείς θα το θέσουμε εκεί όπου η Χούντα της Καστίγια έχει αποφασίσει ότι πρέπει να κατασκευαστεί. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε κύριε Σμέιερ. Κοιτάξτε, έχουμε στην ε, Ολομέλεια πρόσφατα την ψήφιση της έκθεσης Άουκεν ε, που αναφερόταν ε, σε θέματα χωροταξίας και κατασκευών. Η ομάδα μου κατέθεσε μια τροπολογία που εγκρίθηκε ότι στην Ισπανία το μοντέλο της ανάπτυξης ε, και της χορταξίας έχει θίξει άμεσα την ε, πολιτιστική κληρονομιά και υπήρχε αντίκτυπος ε, σε ιστορικές τοποθεσίες ή κοντά σε ιστορικές τοποθεσίες. Αυτό είναι η κοντα σε ιστορικες τοποθεσιες αυτο ειναι η διθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ νομίζω ότι σε μια συγκεκριμένη περίπτωση μπορούμε να μιλήσουμε για ένα έργο αφενός της περιβαλλοντικής πόλης που σαφώς θίγει αυτό που θέλαμε εμείς να πούμε σε αυτή την τροπολογία και αυτό είναι ένα κακό παράδειγμα ε, και εγώ σε ό,τι με αφορά νομίζω ότι το έχουμε ήδη λύσει αυτό το θέμα ε, και πραγματικά ε, εδώ μιλάμε για ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο δεν είναι καθόλου βιώσιμο. Πάντως, ε, αυτή η περιβαλλοντική πτυχή, Πρόεδρε, ε, για αυτή την περιβαλλοντική πτυχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να έχει μία πιο κάθετη και πιο σαφή θέση, πιστεύω εγώ. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι άκουσε πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη ζήτησή μας, τέτοιο ισχύει και με τους αναφέροντες. Έτσι λοιπόν τώρα θα δώσω το λόγο στον ε, αναφέροντα για να μπορεί εσύ να σχολιάσει πολύ σύντομα τα όσα άκουσε, να τονίσετε τα κύρια επιχειρήματα που θέλετε να υποβάλλετε στο τέλος σας παρακαλώ. Η δική μου πρόταση είναι η εξή. Νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την ε, αναφορά και στη συνέχεια να ε, στείλουμε μια επιστολή στον Υπουργό Πολιτισμού στην Ισπανία και να παρουσιάσουμε το θέμα αυτό. Φυσικά θα προωθήσουμε τα επιχειρήματα ε, των αναφερόντων και θα συμπεριλάβουμε και μια σύνοψη της συζήτησης ε, που έγινε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και θα ζητήσουμε να ξεκαθαριστεί το θέμα. αυτήν την η πρότασή μου, αλλά δίνω το λόγο για τρία λεπτά στον αναφέροντα για να κάνει μια σύνοψη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπάμαι που όλα τα εμπλέκουμε. Νομίζω ότι στη φωτογραφία που σας παρουσίασα βλέπετε πως ε, όλα αυτά τα έργα θυγούν άμεσα ή έμεσα μια εμβληματική ιστορική τοποθεσία όπως είναι η Νουμάσια. Αυτό αναφέρομαι και στα δύο έργα και στην περιβαλλοντική ε, πόλη αλλά και στο Σόρια 2 υπόθηκε ότι δεν ε, υπάρχουν ε, καταλογοποιημένες ιστορικές ε, τοποθεσίες. Τώρα όντως δεν υπάρχουν, αλλά η έκθεση αρχαιολογικού αντικτύπου λέει γιατί δεν χρησιμοποιείται να σας πω, ούτε η κλίμακα η κατάλληλη, λέει, και κόβεται το μικρόφωνο της ομιλήτριας, ότι εκεί μπορεί να, ε, ο Σιπίωνας να είχε χτίσει ε, κάποιο πύργο, αλλά στο τέλος λέει η εκθεσή αυτή ότι καθώς υπάρχει τόσο μεγάλη πλάστηση, τίποτα δεν μπορούμε να πούμε, επομένω προτείνεται ότι όταν θα μπουν τα μηχανήματα ε, να να μπουν με μεγάλη προσοχή. Κοιτάξτε, εγώ είμαι αρχαιολόγος, δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι παραδεκτό. Επίσης, ε, αναφερθήκατε ότι οι δύο διαφορετικοί είναι οι Δήμοι της Όρια και του Καρά. Είναι εντάξει, αλλά κοιτάξτε, ε, πριν ε, χίλια χρόνια μιλούσαμε για μια ενιαία περιοχή και εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν τέτοιες διαιρέσεις ότι αυτά πάνε στον ένα Δήμο και τα άλλα στον άλλο ή λέμε τώρα ο ένας Δήμος είναι του ένα κόμματος και ο του άλλου. Εδώ δηλαδή ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλο και δηλαδή αυτό το λέω και αισθάνομαι πραγματικά πάρα πολύ άσχημα. Οι εκπρόσωποι ε, των μεγάλων κομμάτων που θα έπρεπε να υπερασπίζουν κάτι τόσο σημαντικό όπω είναι η νουμάνσια, γιατί δεν είναι εδώ μια οποιαδήποτε τοποθεσία για την οποία μιλάμε. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία πραγματικά έχει επιβιώσει 2.000 χρόνια και έχει διαδραματίσει ρόλο στη ζωγραφική, στη λογοτεχνία. Είναι μια κληρονομιά που οφείλουμε να την προστατεύσουμε και να τη διατηρήσουμε. Αν βρισκόμαστε σε άλλη πόλη, οπωσδήποτε θα είχε κηρυχθεί ε, πολιτιστική κληρονομιά τη ανθρωπότητα, παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Έτσι νομίζω ότι εδώ είναι λυπηρό που έρχομαι να υπερασπίσω τα προφανή, αλλά τέλο πάντων σα το αφήνω να το σκεφτείτε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε την πρότασή μου. Νομίζω ότι αυτή θα ήταν η καλύτερη λύση σε αυτό το στάδιο και ελπίζω να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. αφού Θα έχουμε λάβει και τις απαραίτητες πληροφορίες από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μάλιστα, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Να δηλώσω ότι εγώ διαφωνώ με όσα είπε η κυρία Πέρεξ και αν η ίδια είχε δράσει στο Πανεπιστήμιο, εγώ ήμουν πρόεδρο της Υποεπιτροπής τη Πολιτική Κληρονομιά του Συμβουλίου τη Ευρώπη, και μιλάμε για Ευρώπη που φτάνει από τον Ατλαντικό ω τα Ουράλια. Ζω σε μια πόλη η οποία είναι παγκόσμια υποστηρική κληρονομιά και πραγματικά σέβομαι ε, την κληρονομιά στην Ουμάντσια και από την αρχή μέχρι τώρα που ξεκαθαρίζει το θέμα ε, είδαμε ένα το revolutum και μπλέξαμε το έργο ε, Σόρια 2 με το έργο της περιβαλλοντικής πόλης. Εγώ απλώς ήθελα να ξεκαθαρίσουμε και να διαφοροποιήσουμε το ένα από το άλλο. Επίσης, εδώ εκπρόσωπο από ε, την κοινωνία των πολιτών. Μάλλον βλέπω ότι είναι πάρα πολύ καλό και συμφωνώ η κοινωνία των πολιτών να μας ε, καταθέτει την άποψή της. Ε, όμως δεν μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι εδώ εγώ δεν έρχομαι να υπερασπίσω την πολιτιστική οικονομία της Νουμάνσια. Μάλιστα, κοιτάξτε, ε, εσείς δεν αναφερθήκατε, δεν έφερατε κάποια αντίδραση στην την πρόταση. Θα γράψω στον Υπουργό Πολιτισμού, θα ζητήσω εξήγησεις και θα επανέλθουμε. Εγώ νόμιζα γι' αυτό είχα ζητήσει το λόγο για να σχολιάσετε την δική μου πρόταση, αλλά αναφερθήκατε σε κάτι άλλο. Ας προχωρήσουμε τώρα στο σημείο 21 αναφορά 587-2008 του κυρίου Χωσελουίνες Φερνάντες ε, Φουέρος. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ε, Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ εκπροσωπώ, θα δώσω το λόγο στην πρόεδρο της ε, Ένωσης ε, Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε και πάλι την ευκαιρία να εκφράσουμε εδώ τα επιχειρήματά μας. Ε, ε, η αποδοχή που δείχνει αυτός ο οργανισμός απέναντι στο θέμα αυτό έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τον επιφανειακό χαρακτήρα και την απογοητευτική απάντηση μέσω της ΓΔ περιβάλλοντος. Η απάντηση αυτή ε, πραγματικά καταρρύπτεται βάσει των εγγράφων που παρουσιάζουμε εμείς σύμφωνα με ε, τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Οι κυβερνήσεις Ισπανίας και καθορίζουν ότι το Ίδρυμα Ψερβατόριο Πορτο δημιουργήθηκε για να εγγυηθεί την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των αντισταθμιστικών και διορθωτικών μέτρων. Επομένως, μας εκπλήσει ότι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 πρώτη ενέργεια αυτής της ήταν ε, να προσπαθήσει να ελέγξει και να προωθήσει μια έκθεση που θα επέτρεπε την ε, μη προστασία ενός από τα είδη που συμπεριλαμβάνονταν στον κατάλογο των απειλούμενων ειδών των Καναρίων, καθώς ε, και την οδηγία οικοτόπων για της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να αποφευχθεί η κατασκευή αυτής της υποδομής να μετατραπεί σε οικολογικό έγκλημα. Η επιστημονική κοινότητα των δύο πανεπιστημίων των ίσων ε, των Καναρίων ε, ε, απαντά με πυγμή κατά αυτής της έκθεσης επίσης σε αυτή αυτό το παράπτωμα αναφέρεται το ανώτερο κέντρο επιστημονικών ερευνών και το αυτόνομο πανεπιστημίο της Μαδρίτης και γνωστοποιούν στο Υπουργείο ε, Περιβάλλοντος ε, την κάθετη απόρριψή τους. Η στάση της επιστημονικής κοιμότητας ε, δείχνει την ε, μεροληψία του Ιδρύματος Οψερβατόριου Πόρτο των στην πολιτική εξουσία. Αυτή η απάντηση ε, επίσης συνοδεύτηκε με μια μεγάλη διαδήλωση στις 14 Μαρτίου όπου συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι και διάφορες ε, συλλογικότητες επιστημονική απάτη προστίθεται και η χειραγώγηση της διοικητικής διαδικασίας, του να αφαιρεθεί από τον ε, κατάλογο ε, αυτών των στοιχείων. Οι κύριες οικολογικές οργανώσεις της Ευρώπης ε, τονίζουν στο μάλλον ε, παρακαλούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος να ε, ακυρώσει την δήλωση περιβαλλοντικού αντικτύπου του σχεδίου. Επίσης και το Σοσιαλιστικό Κόμμα απαιτεί να γίνει μια νέα μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Το σχέδιο του λιμάνιου της Γραναδίγια έχει ε, ένα δυστυχές προηγούμενο, το λιμένα του Αρινάγα στις Πάλμας Δεγκράν Κατήρε και το οποίο τρία έτη αφού ολοκληρώθηκαν ε, οι εργασίες παραμένει ανενεργό. Ε, αυτό έχει να κάνει με τους ανέμους που φυσάνε και πραγματικά έχουν ως αντίκτυπο να είναι αδύνατο να ε, αγκυροβολήσουν ε, τα πλοία και να φορτώσουν ε, και να ξεφορτώσουν. Επίσης, μία ακόμη ομοιότητα έχει να κάνει με την αποψήλωση ουσιαστικά των διαρθρωτικών κονδυλίων και τον περιβαλλοντικό αντίκτυμο που θα είχε η κατασκευή του λιμένα της Γραναδίγιο. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος απάντησε ότι δεν έχει λόγους για να θεσπιτήσει την μεροληψία του Ιδρύματος, όμως τόσο σας ανέφερα εδώ, δείχνουν ακριβώς τη δική μας καταγγελία θα μπορούσε να αποτελεί κάλλιστα μέρος της έκθεσης Άουκεν που πραγματικά αμφισβήτησε την περιβαλλοντική και χορταξική διαχείριση της Ισπανικής ακτής. Για όλα αυτά ζητάμε στην Επιτροπή αυτή τα δύο τεινά. Να ε, διορίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων που να μελετήσει και να αναλύσει την ε, οικονομική περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την επιχειρησιακή βιωσιμότητα και να καλέσει τα μέρη να συνδυάσουν προκειμένου να αναλύσουν τα υπέρ και τα κατά αυτής υποδομής. Δεύτερον, να ζητήσει από την Επιτροπή Περιβάλλοντος να θεωρήσει την ε, έκθεση που ήταν, ε, υλοποιήθηκε το 2006 και ήταν ε, ευνοϊκή, καθώς ε, οι αναφέροντες καταγγέλουν ότι αυτές οι πληροφορίες που είχαν χορηγηθεί από τις Ισπανικές Αρχές και σε οποίες βασίστηκε η απόφαση της Επιτροπής είναι ψευδείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το, λόγο στον πρόσωπο της Κομισιόν. Θα μιλήσω εξ ονόματος ε, της ε, ΓΑΜΑΔΑΛΙΤΑ Περιβάλλοντος, Πρόεδρε. Καταρχήν, να επισημάνω ότι το αντικείμενο αυτής της αναφοράς ε, ήταν η αμεροληψία ε, του Παγκοσμίου Ιδρύματος ε, του παρετηρίου, του Λιμένα της Γραναδία και των όσων εκπροσωπούν τις ενώσεις για την περιβαλλοντική πτυχή. Αυτό ήταν το αρχικό αντικείμενο της αναφοράς που έγινε σε αυτήν την Επιτροπή και για την αναφορά αυτή η Κομισιόν έχει γνωστοποιήσει το εξή. Η Κομισιόν πολλές φορές τράφηκε στι ισπανικέ αρχές για την περίπτωση του λιμένα της Γραναδίγια και δύο φορές στις Ισπανικές αρχές ζητώντας διευκρινήσεις για τις διαδικασίες εξέτασης που έγιναν σε ό,τι αφορά τη δράση ε, των ε, συμμετεχόντων ε, από τους εργοδότες. Επίσης, ε, ε, ζητήθηκαν εξηγήσεις γιατί επιλέχθηκε αυτή η τοποθεσία και οι Ισπανικές αρχές αναφέρθηκαν στο 3-2 στο διάταγμα 123. η Επιτροπή πιστεύει ότι αυτή αποτελεί μια δημόσια ανοιχτή διαδικασία και σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από τις Ισπανικές Αρχές η διαδικασία επιλογής ε, ε, έγινε βάση της νομοθεσίας ε, και οι υποψηφιότητες ε, δηλώθηκαν σε δύο τοπικές εφημερίδες αλλά και στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης των Καναρίων. Παράλληλο το ότι μόνο μία περιβαλλοντική οργάνωση παρουσίασε την υποψηφιότητά της, η Κομισιόν θεωρεί ότι η νομική διαδικασία, κατά την νομική διαδικασία δεν υπήρχε παραβίαση. Ο κύριος Leclerc. Μάλιστα. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν αυτά που θα σας πω ξεπεράσουν το αυστηρά πλαίσια της αναφοράς που είναι ένα θέμα περιβάλλοντος. Εγώ εκπροσωπώ τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής που διαχειρίζεται τα διαρθρωτικά ταμεία και στα Καναρίους. Λοιπόν, το κατά πόσον είμαι αρμόδιος ή όχι και σε τι βαθμό ε, και το κατά πόσον το λιμάνι της Γρεναδούλας έχει χρηματοδοτηθεί νομοτύπως αφορά το εξής θέμα. Η κατασκευή του νέου λιμανιού της Γρεναδούλας εμφαίνεται στον κατάλογο τοποθεσιών που μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν με βάση ένα πρόγραμμα ΦΕΝΤΕΡ και Ταμείου Συνοχής 2007-2013 και τα σχέδια που έχουν εκεί υποβληθεί θεωρούνται κατάλληλα για συγχρηματοδότηση από το 2007 και μετά. Τώρα για να συγχρηματοδοτηθούν όμως επειδή πρόκειται για μεγάλα προγράμματα πρέπει να υπάρξει απόφαση μεμονωμένη για το καθένα της Κομισιόν. Όχι μόνο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής αλλά όλων των αρμοδίων υπηρεσιών, περιβάλλοντος και μεταφορών κλπ. Μέχρι τώρα, άρα δηλαδή χρειάζεται τα κράτη-μέλη να κάνουν, να υποβάλουν αίτηση συγχρηματοδότησης. Η αίτηση αυτή μας ήρθε την περασμένη εβδομάδα αλλά βέβαια είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε ότι μπορούμε να πάρουμε και απόφαση για την συγχρηματοδότηση του προγράμματος αυτού από το ΦΕΝΤΕΡ. Πρέπει πρώτα να τη μελετήσουμε και να δούμε τα, τις λεπτομέρειες. Δεν έχουμε τελειώσει λοιπόν ακόμα και γι' αυτό μπορώ να δηλώσω ότι μέχρι τώρα δεν έχει χορηγηθεί καμία χρηματοδότηση από το λιμάνι της Γραναδούλας από κανένα ταμείο, ιδίω συνοχή. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα διαβάσω τον κατάλογο των ομιλητών και έτσι θα αλήξει ο κατάλογος αυτός. Μέιερ, Κάσμαν, Αν θέλει κανείς άλλος να λάβει το λόγο να το πει τώρα, γιατί θα κλείσω τον κατάλογο. Λίγη κλείνει ο κατάλογος. Έκλεισε. Δύο λεπτά ο κάθε ομιλητής και η κάθε ομιλήτρια. Ο κύριος Μεδίνος. Πρόεδρε. Μεταξύ της τεκμηρίωσης ε, που παρουσίασαν ε, οι αναφέροντες έχουμε και μία πράξη του Δικαστηρίου των Κανονιών 13 Μαρτίου και με την πράξη αυτή αναστείλεται η εξέταση των διαδικασιών για την ε, καταλογοποίηση και μιλάμε για ουσιαστικά ένα ε, ε, ένα, μια απόφαση που σημαίνει, μάλλον μια πράξη που σημαίνει ότι μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα πρέπει να τοποθετηθεί το δικαστήριο. Έτσι λοιπόν, καθώς εκκρεμεί μια δικαστική απόφαση, θεωρώ ότι ε, εμείς πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό σε σχέση με τη διαδικασία. Εγώ δεν λέω ούτε να συνεχιστεί, ούτε να σταματήσει, αλλά ε, ουσιαστικά να περιμένουμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου, γιατί εκεί θα καθορίζονται ε, πτυχές όπως είναι οι εθνικές αρμοδιότητες, ε, το θέμα της ε, αναλογικότητας κτλ. Έτσι λοιπόν η πρότασή μου είναι πολύ συγκεκριμένη, δηλαδή το θέμα που υπάρχει επιτάπητος, να το κρατήσουμε επιτάπητος μέχρι να έχουμε την οριστική απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου των Καναρίων. Κύριε Τουρκάη, για δύο λεπτά. Άκουσα τον σύντροφο Μεδίνα και θα ήθελα και εγώ στην παρέμβασή μου να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Μεδίνα. Όπως είπε, πρέπει να λάβει το του δικαστήριο την απόφαση αυτή. Και κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι έχουμε δει κι άλλες φορές ε, εδώ στην Επιτροπή μας τέτοιες αναφορές ε, ε, τις ε, οποίες ουσιαστικά τις παγώναμε μέχρι να υπάρχει η δικαστική απόφαση και εγώ θα ήθελα να εθετήσουμε αυτό το μέτρο και να ζητήσω να αναστείλουμε τη συζήτηση για αυτή τη αναφορά μέχρι να έχουμε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστήριου κ. Μέγερ. Ναι, νομίζω ότι είναι προφανές ότι αυτή η αναφορά θα πρέπει να μείνει ανοιχτή, ζωντανή, γιατί έχουμε ε, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που έχουν ληφθεί από το δικαστήριο έτσι ώστε να σταματήσει ένα έργο που το 2006 η Κομισιόν το είχε κρίνει καλό. Έτσι λοιπόν ε, υποχρεούμαστε να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αίτηση. Νομίζω ότι αυτή είναι η θέση μου για το θέμα ε, νομίζω ότι τη της πρέπει να αναθεωρήσει η Κομισιόν ε, τη θέση που έλαβε το 2006. Γιατί κοιτάξτε, εδώ το δικαστήριο, και μιλάμε για το νότο το δικαστήριο των Κανερίων και λαμβάνει ε, τέτοια ε, μέτρα ασφαλιστικά για να θέσει τέλος στο έργο και μάλιστα λαμβάνει υπόψη και την επιστημονική γνωμοδότηση του ανώτερου επιστημονικού οργάνου της Ισπανίας. Αυτό σημαίνει ότι η κατασκευή ενός μέρους του λιμένα είναι απόλυτα αυθαίρετη γιατί εδώ πρέπει να δούμε και τι συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των ειδών που απειλούνται. Έτσι λοιπόν, εγώ συμφωνώ με τους ε, συναδέλφους που είπαν ότι πρέπει να μείνει ανεκτό αυτό το θέμα, αλλά θέλω να πω και στην Κομισιόν να αναθεωρήσει τη θέση της του 2006, γιατί υπάρχουν εναλλακτικέ και γιατί η κοινή γνώμη είναι εντελώς κατά. Και είδατε ότι πολύ πρόσφατα έλαβε χώρα μια πολύ μεγάλη διαδήλωση σχετικά. Ευχαριστώ, κύριος Χάμερστάιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ κρίμα που οι δύο μεγάλες ομάδες δεν μας άφησαν να επισκεφτούμε την περιοχή της Γραναδία γιατί εκεί ε, έχουμε ε, μια από τις μεγαλύτερες ε, κοινωνικοπολιτικέ διαμάχες που υπάρχουν στην Ισπανία. Και είναι κρίμα που πραγματικά εξευτελίστηκε τόσο πολύ κομισιόν, θα έλεγα εγώ, γιατί φαίνεται ότι ένας δικαστής στην Τενερίφη μπορεί καλύτερα να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό δίκαιο. Mm. Και μάλιστα φαίνεται ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να το πράξει και υποχωρεί, ε, υποχώρησε πριν δύο χρόνια ενώπιον πίεση των δύο μεγάλων κομμάτων. Γιατί υπάρχουν πληροφορίε που αιτιολογούν να ξανανοίξει αυτό το θέμα από την Κομισιόν. Καταρχήν, Έχουμε αυτή την ε, αναστολή, τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά στην Ισπανία, γιατί η απόφαση, σύμφωνα με την απόφαση, έχουμε αναπόδραστες ε, επιπτώσεις ε, στον βυθό. Και ξέρουμε ότι αυτή την επιστημονική γνωμοδότηση την εκπώνησε το Πανεπιστήμιο. Και επίσης και δέχουμε και δεύτερη μελέτη που δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο. Αυτή είναι νέα μελέτη που είδαμε σήμερα το πρωί και προέρχεται από ένα καθηγητή ε, αρμόδιο για τη θαλάσσια κυκλοφορία και λέει ότι αυτός ο λιμένας δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω των ανέμων που φυσάνε εκεί. Και υπογράφεται αυτό από τους ε, διασημότερους καθηγητές ε, της Ισπανία, Γιατί λοιπόν θέλετε να χρηματοδοτήσετε ένα λιμένα που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, που δεν χρησιμεύει σε τίποτα, αυτό να το θέσω στον κύριο Λεκλέρκ της περιφερειακής πολιτικής. Και αν είναι αλήθεια ότι ένα αυτό το λιμάνι δεν μπορεί να λειτουργεί 180 μέρες το χρόνο λόγω των ισχυρών ανέμων, ε, τότε γιατί να χρηματοδοτηθεί αυτό το σχέδιο από ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ενώπιον ε, των εργών, ε, μπροστά από τα έργα που έχουν ξεκινήσει, υπάρχει μια μεγάλη αφήσα πολύ, συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι νόμιμη ε, αυτή η πινακίδα. Η κυβέρνηση των Καναρίων δήλωσε ότι λαμβάνει 68 δισεκατομμύρια ευρώ για τα έργα αυτά. Εμεί τώρα ακούσαμε ότι δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση, ούτε καν έχει ζητηθεί. Είναι νόμιμο δηλαδή η κυβέρνηση εκεί στα Κανάρια να θέτει αυτή την πινακίδα και μάλιστα ε, να ε, στέλνει και άρθρο στον τύπο που να λέει ότι έχει ζητήσει τέτοια χρηματοδότηση τι μας ε, λέει η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής ε, για αυτή τη δημόσια δήλωση, γιατί είναι σημαντικό. Γιατί ε, το κύριο επιχείρημα της κυβέρνησης των Καναρίων κατά του να ανασταλούν οι εργασίες είναι ότι δεν θα μπορούσαν να απορροφηθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουν δοθεί. Και επομένως, αν αυτό αποτελεί, έχει ουσιαστική σημασία για τη λήψη της απόφασης από το δικαστήριο, πρέπει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γίνεται με τα κονδύλια αυτά. Πρέπει οπωσδήποτε να δοθούν για αυτό το λιμένα στην Κραναδία ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για κάτι άλλο. Και επίσης το κοινωνικό στόχος ε, ενός ε, έργου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Εδώ δεν είναι σαφές αυτός ο στόχος. Η κυβέρνηση των Καναρίων μας λέει ότι υπάρχει έλλειψη δυνατότητας να διευρυνθεί ο λιμένα Σαντακρούν. Και, ε, Αυτές ήταν ε, πληροφορίες ε, που δεν ήταν σωστές, σύμφωνα με πολλούς εμπειρογνώμονες και θέλουμε να ξέρουμε αν η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος έχει αμφιβολίες για τις ε, πληροφορίες που έχουν στείλει οι αρμόδιες ισπανικές αρχές. Μα έχω διαδικαστικό. Α, διαδικαστικό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, καθώ είναι ένα διαδικαστικό θέμα. Δεν έχω τίποτα κατά του Μάικλ. Το αντίθετο, μάλιστα, αλλά εδώ μιλάμε για μία αναφορά η οποία θέτει ένα ζήτημα. Δεν μπορούμε να ερχόμαστε εδώ να ζητάμε εξηγήσει για αυτό το σημείο, για το τι λέει την ακίδα ή για άλλο θέμα, γιατί διαφορετικά τι θα κάνουμε. Κοιτάξτε, ήδη έχει συζητηθεί αυτό το θέμα. Εδώ έχουμε μια αναφορά για την ανεξαρτησία του ιδρύματος αυτού του δημοσίου. Ας μιλήσουμε γι' αυτό, όχι για πινακίδες, γιατί ε, αν ξαναμιλήσουμε για το ελληνικό της δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο, ήδη το συζητήσαμε αυτό το θέμα και ήδη έχουμε αποφασίσει. Κύριος Χάμερστάιν. Πρόεδρος διακόπτη, συγγνώμη. Όταν ε, κάποιος έχει χρόνο ομιλίας, μπορεί να λάβει το λόγο το άτομο αυτό και να πει ό,τι θέλει μπορεί να αναφερθεί συγκεκριμένα. Uh, Για το διάλογο είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει παρέμβαση κτλ. Αλλά είναι φανερό ότι ο κ. Μεδίνα έχει απόλυτο δίκιο. Το θέμα το χειρίζεται το δικαστήριο. Δεν πρέπει να προδικάσουμε τίποτα. Αλλά να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά και γιατί τίθεται το θέμα νέας περιβαλλοντολογικής αξιολόγησης πιθανής. Να μην προδικάσουμε λοιπόν. Συμφωνώ βέβαια με τους αναφέροντες και τους υποστηρίζω αλλά πρέπει να περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε πολλά ερωτήματα προς την Κομισιόν. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να τις προτείνω να απαντήσει στα ερωτήματα, μόνο αυτό, όχι να θίξει γενικότερα το θέμα, μόνο τα ερωτήματα. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Έμαθα ότι θα γινόταν η συνεδρίαση αυτή πολύ λίγο πριν έρθω και γι' αυτό νομίζω ότι, γι' αυτό νομίζω, ε, νομίζω όμως ότι καλά έκανα που ήρθα γιατί τα ερωτήματα αυτά και που μάλιστα αφορούν την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής είναι αυτά που σας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, πολλά ερωτήματα τέθηκαν. Αν κατάλαβα καλά αυτά που είπε ο κύριος Χάμερστάιν, είπε ότι η Κομισιόν θα συγχρηματοδοτήσει το λιμάνι αυτό. Όχι. Θα δούμε αν θα συγχρηματοδοτήσει σύμφωνα με την ενομισμένη διαδικασία. Δεν προδικάζουμε το αποτέλεσμα της εξέτασής μας. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα καταλήξει σε αποδοχή της χρηματοδότησης. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Οι νέες μελέτες που υποβλήθηκαν, εμείς δεν τις ξέρουμε, δεν τις λάβαμε. Φαίνεται ότι μία αφορά την μη λειτουργικότητα του λιμανιού αυτού ε, τέτοιου είδους μελέτες προφανώς πρέπει να τις δούμε, θα τις λάβουμε σοβαρά υπόψη όταν εξετάσουμε αυτή την αίτηση συγχρηματοδότησης, όπως και όλα τα άλλα στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να κρίνουμε κατά πόσον γίνεται αποδεκτή. Για το θέμα τώρα του πανό ή της πινακίδας. Είδα και χθες φωτογραφίες της που έλεγαν ότι το λιμάνι της Γρεναδούλας εστάκο φινανσιάδο, δηλαδή συγχρηματοδοτείται ήδη. Έλεγε και το ποσοστό της συγχρηματοδότησης. Αυτά δεν είναι Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι όπως είπα και προηγουμένως, το σχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνεται στον ενδεικτικό πίνακα προγραμμάτων που μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Συνοχής και το ΦΕΝΤΕΡ 2007-2013 οι δαπάνες που προβλέπει μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από το 2007 και μετά και το κράτος μέλος που ενδιαφέρεται έχει την υποχρέωση κανονικά να βάζει μια πινακίδα που να γράφει την ενωσιακή συγχρηματοδότηση σε κάθε έργο που συγχρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία. Το πρόβλημα είναι ότι η διατύπωση της πινακίδας αυτής είναι λανθασμένη. Λέει ότι ήδη συγχρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία και αυτό μπορεί να οδηγήσει πολλούς σε λάθη και παρεξηγήσεις. Διότι δεν έχει ακόμη ληφθεί καμία απόφαση από την Κομισιόν αποδοχής της συγχρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία και γι' αυτό δεν, η διατύπωση αυτή είναι υπερβολική. Δεν μπορούμε όμως και να πούμε ότι παρανόμησε το κράτος μέλος αφού ο κανονισμός για την πληροφόρηση ως προς τα προγράμματα προβλέπει μια τέτοια πινακίδα. Δεν έκανε και καμία παραβίαση αλλά να υπερέβαλε πώ να το πω. Γενικά μάλιστα εμείς προσφεύγουμε όταν δεν βάζουν τις πινακίδες στα κράτη μέλη. Ε, ναι, έτσι είναι δυνατά. Στα έργα που συγχρηματοδοτούνται. Και αφού τελειώσουν. Αυτά είχα να σας πω. Κοιτάξτε κυρίες και κύριοι. Αφού συμφωνούμε οι περισσότεροι να την αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και αφού το δεύτερο επιχείρημα του κυρίου Μεδίνα και άλλων είναι επίσης να περιμένουμε για να λήξει η διακαστική διαδικασία στην Ισπανία, προφανώς θα περιμείνουμε. Αλλά θέλω επίσης να, ρωτήσω την, να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα όσα μας είπε και ό, μερικά που δεν μας είπε γιατί είπατε ότι μάθατε πολύ αργά ότι θα γινόταν η συνεδρίαση αυτή και δεν είστε προετοιμασμένος καταλήλως. Δεν φταίμε εμείς βέβαια γι' αυτό, γιατί εμείς γνωστοποιήσαμε γέρος. Αλλά τέλος πάντων, όλα όσα είπατε και αυτά που δεν μπορούσατε να πείτε γιατί δεν είστε ο πιο αρμόδιος, να μας τα γράψετε και όλα να τα γράψετε και τους πίνακες. Τελειώνει και αυτό λοιπόν το θέμα και πάμε τώρα στο 22, αναφορά 554 του 2006. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν πρώτα, Καβέσινα Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτή η αναφορά αφορά έναν αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας Ο, μικ... ο πρόεδρος μιλάει χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπα, αυτή η αναφορά αφορά την κατασκευή, το σχέδιο κατασκευής ενός αυτοκινητοδρόμου ταχείας κυκλοφορίας που θα διασχίζει το κέντρο της Γκλίβιτσε. Έχει χωριστεί σε τέσσερα επιμέρους τμήματα η κατασκευή αυτού του αυτοκινητοδρόμου και αποτελεί αντικείμενο μιας ενιαίας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η Επιτροπή, η Κομισιόν έχει κάνει μια σχετική ε, μελέτη και έχει παρουσιάσει τα αποτελέσματα στις ε, πολωνικές αρχές. Οι πολωνικές αρχές με τη σειρά τους όφυλαν να εκπονήσουν μια επίσης ενιαία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλα τα επιμέρους τμήματα του αυτοκινητοδρόμου οι πολωνικές αρχές επίσης ανέλαβαν να διασφαλίσουν ότι αυτή η μελέτη θα, ήταν, θα, θα συμμορφωνόταν με όλες τις, ε, όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ως τον Οκτώβριο του 2009 έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η σχετική έκθεση. Μετά την ολοκλήρωσή της, οι επενδυτές, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα κατέθεταν τη, τα αιτήματά τους. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα συμπεριλάβει και μια δημόσια διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις πληροφορίες, αυτά τα δεδομένα, προφανώς η Κομισιόν δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα Γι' αυτό και η Κομισιόν συνιστά την περάτωση, το κλείσιμο αυτής της αναφοράς. Αν κάποια στιγμή ο αναφέρον θεωρήσει ότι πρέπει να τεθεί ένα αμφιβόλο η, η σωστή διεξαγωγή της ε, διαδικασίας, η Επιτροπή, η Κομισιόν ευχαρίστως να ξανανοίξει την ε, υπόθεση. Επί του παρόντος πάντως δεν υπάρχουν στοιχεία που να μας επιτρέπουν να πούμε ότι έχει υπάρξει παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι με αυτά που άκουσα γιατί η αναφορά βασίζεται, ενέχει, περιέχει μια παρεξήγηση. Καταρχάς πρέπει να γνωρίζουμε ότι πρέπει να, να γνωρίσουμε τις συγκεκριμένες συνθήκες της κατασκευής αυτής. Ο αυτοκινητόδρομος αυτός θα, θα διέρχεται από 14 δήμους. Σε, ορισμένες... σε ορισμένα σημεία θα, ο δρόμος θα διέρχεται από το κέντρο των πόλεων σε άλλα όχι. Η αναφορά που εξετάζουμε έχει, δεν έχει έγκυρη νομική βάση γιατί το νομικό καθεστώς έχει στο μεταξύ μεταβληθεί. Οπότε είναι πραγματικά πρόωρο και όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν δεν έχουν, γίνει, δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα στάδια όπως θα έπρεπε. Οπότε θα θέλαμε μερικές ε, διευκρινήσεις ως προς την κατάσταση από νομικής άποψης. Όσον αφορά την περιβαλλοντική πτυχή, υπάρχουν επίσης αμφιβολίες και ενδεχομένως παρεξηγήσεις, αλλά αξίζει τον κόπο να ακούσουμε παραπάνω. Πρόκειται για αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας, expressway, όχι highway, και η εκπομπή αέριων ρήπων είναι περισσότερο πρόβλημα στις χαμηλές ταχύτητες και όχι στις υψηλές. Όταν η το όριο ταχύτητας είναι 70 χιλιόμετρα την ώρα, Οπότε οι εκπομπές δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλές. Τα μνημεία που υπάρχουν στην πόλη της Γκλιβίτσα δεν θα υποστούν αρνητικές ε, συνέπειες. Το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου που θα διέρχεται από την κατοικημένη ζώνη θα, δεν θα είναι ανοιχτό. Θα κατασκευαστεί μια σύραγγα, οπότε οι εκπομπές δεν θα αυξηθούν στη γύρω περιοχή ίσως και να μειωθούν. Γιατί στην πόλη της Γκλιβίτσε είναι καθημερινό φαινόμενο τα μποτιλιαρίσματα. Η διέλευση των φορτηγών ε, αποκλείει την... προκαλεί μάλλον προβλήματα συμφόρησης στους δρόμους. Οπότε μετά την ολοκλήρωση, μετά την κατασκευή της σύραγγας, είναι λογικό να αναμένει κανείς ότι οι εκπομπές θα μειωθούν και θα αμπληθεί και το πρόβλημα το, της συμφόρησης. Είναι όσον αφορά τώρα το, τους ε, υδάτινους πόρους, την, τον υγροφόρο ορίζοντα, επίσης δεν αναμένουμε αρνητικά αποτελέσματα. Οι ροές των, οι υδάτινες ροές δεν, τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν σαν βάση τις υδάτινες ροές δεν, είναι, δεν έχουν βάση στην πραγματικότητα. Η πυκνότητα της κυκλοφορίας θα μειωθεί σε, στο τμήμα που μας ενδιαφέρει. Άρα ξανά οι εκπομπές ε, αναμένεται να μην είναι υψηλέ. Οπότε πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να κλείσει το θέμα. Πολύ σύντομα, άκουσα όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Εμείς από την πλευρά μας νομίζω ότι, είναι κατάλληλη στιγμή να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς. δεν έχει δοθεί ακόμη σχετική περιβαλλοντική άδεια, αναπτυξιακή άδεια. Οπότε, αν ο αναφέρον μας αποδείξει ότι έχει δοθεί σχετική έγκριση, ευχαρίστως να ασχοληθούμε με το θέμα σε δεύτερο χρόνο. Μπορεί να υποβάλει εκ νέου την αναφορά και να ξαναανοίξει η ίδια αναφορά. Ευχαριστώ, Μάικλ και κύριε Ροσκόφσκι. Οπότε, όντως, είναι η καλύτερη λύση να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς. Η Είμαι υπέρ ε, της περάτωσης σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλω πραγματικά να δώσουμε, να προετοιμάσουμε το έδαφος για εκ νέου εξέταση. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό να ενθαρρύνουμε τον αναφέροντα να την υποβάλει εκ νέου. Ο στόχος είναι να ικανοποιηθούν όσο γίνεται και οι δύο πλευρές. Από ό,τι βλέπω έχει ήδη ληφθεί η απόφαση. Το σημείο 23 έχει μετακινηθεί, οπότε περνούμε στο σημείο 24, αναφορά 480 κάθετος 2007. Θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Πρόκειται για διαδικαστικό θέμα. Όσον αφορά τον κύριο Άτκινς και την sera communiqué aux membres de la Commission ce soir par email. Το σημείο 17 που συζητήθηκε στις 11 Δευτέρου. Ο κύριος Πέτερ Κόλλερ για την επόμενη αναφορά. Σημείο 24. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η αναφορά αφορά ένα, ένα έργο πολεοδομικό έργο, κατασκευαστικό έργο, ο αναφέρον υποστηρίζει ότι το σχέδιο αυτό θα έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, σοβαρές, και ότι πρέπει να γίνει μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από το στάδιο της ε, διαβούλευσης. Μετά τις ε, έως τώρα απαντήσεις στην αναφορά αυτή, η Κομισιόν έκρινε ότι υπό τις ε, συνθήκες που περιγράφονται στην αναφορά έπρεπε να τεθεί το θέμα στις Μαλτέζικες Αρχές, όπως και συνέβη. Μας παρασχέθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις. Οι Μαλτέζικες αρχές ε, μας εξήγησαν ότι το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο προβλέπει την, ε, την κατεδάφιση των υπαρχόντων κτηρίων. Στο, με την σχετική έγκριση των αρμόδιων αρχών η, στην ουσία μόνο το δεύτερο στάδιο, η δεύτερη φάση των εργασιών θα είχε επιπτώσεις για αρνητικές για το περιβάλλον. Διεξήχθη λοιπόν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ειδικά για τη δεύτερη φάση του έργου. Οι Μαλτέζικες Αρχές επίσης μας ανέφεραν ότι η άδεια για την πρώτη φάση δόθηκε στις 25 Ιουλίου του 2006 ενώ για τη δεύτερη φάση στις 6 Ιουνίου του περασμένου έτους οι δύο φάσεις είναι διακριτές λόγω του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ τους. Έγιναν, ε, εξετάστηκαν διάφορες ε, καταγγελίες όσον αφορά την ε, εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και την ε, διεξαγωγή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τη σχετική οδηγία. Η Επιτροπή η Κομισιόν δεν διαπιστώνει παραβίαση της οδηγίας EIA. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλα σχόλια. Αν όχι, να κλείσουμε. Λοιπόν, περατώσαμε και αυτό το σημείο. Περνάμε στο σημείο 25 που έχει να κάνει με τις βελτιστικές πρακτικές. Sir Robert wants to introduce it, but no, to w takim razie odkładamy to na. Κοιτάξτε, να το εισαγάγουμε δεν ξέρω αν θα πρέπει να το συζητήσουμε τώρα κάποια άλλη φορά, γιατί ε, εδώ μπλέκεται και το ΕΛΚ. For mig har det været en vigtig grund til, at jeg også har de punkter, fordi jeg Κοιτάξτε, εγώ ανησυχούσα πάρα πολύ όταν είδα ότι υπήρχε η πρόταση αυτή, γιατί αυτή η πρόταση που αφορά τα ταξίδια με ανησυχεί. Γιατί αν περάσει τότε ε, δεν θα έχει νόημα η Επιτροπή μας. Ίσως ε, θα πρέπει να αλλάξουμε μέχρι και το όνομα για την επόμενη θητεία. Τη στιγμή των εκλογών ε, έχετε μία επιτροπή που είναι κοντά στους πολίτες και που έχει τη δυνατότητα να παρέμβει να μπορεί να δεκπεραιώνει με σοβαρό τρόπο τις ε, καταγγελίες τους, τα παραπονά τους. Αυτό αφενός από την άλλη έχουμε και το πρόβλημα ότι δεν μπορούμε όλοι να, το, ε, να εκφραζόμαστε όσο θέλουμε. Συγγνώμη. Ο Σερ Ρόμπερτ δεν είναι εδώ, επομένως προτείναμε να αναβάλουμε το θέμα μέχρι την επόμενη συνάντηση. Πρόεδρε, δεν θέλω να διακόψω την κυρία Άουκεν. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό προς το πρόσωπό της, αλλά δεν νομίζω ότι είναι λογικό ένα τόσο σημαντικό θέμα να το βάζουμε στην ημερησία διάταξη στο τέλο του απογεύματος, γιατί υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις στις πολιτικές ομάδες, ε, και δεν έχουμε μόνο δύο πολιτικές ομάδες σε αυτήν την Επιτροπή, υπάρχουν πολλές πολιτικές ομάδες και θα ήθελα να ακούσω και τη δική τους άποψη. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι δεν θα ήταν κατάλληλο να συνεχίσουμε τώρα αυτή τη συζήτηση χωρίς ε, μάλιστα να υπάρχει και ο συντονιστής ε, εδώ του ΕΛΚ για να παρουσιάσει το σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Μάλιστα. Κυρίε και κύριοι, εγώ ήθελα να υποστηρίξω τον κύριο Κάσμαν για την ε, αναβολή αυτή. Μάλιστα, ευχαριστώ. Πρόεδρε, μία διευκρίνηση, κυρία Λέια. Τα κείμενα που έχουμε εδώ, που μας έχετε διανύμει, στην ισπανική εκδοχή υπάρχει μία πρόταση, ενώ στη συνέχεια στην ε, γνωμοδότηση υπάρχει ένα τροποποιημένο κείμενο στα αγγλικά. Μήπω υπάρχει αυτό το κείμενο και στα ισπανικά, αυτό το τροποποιημένο κείμενο. Γιατί έχουμε δύο κείμενα, δηλαδή ένα στα ισπανικά και ένα στα αγγλικά. Απλώς για να ξέρω όταν το συζητήσουμε, αν θα πρέπει να έχω και τα δύο κείμενα στα ισπανικά. Αν αναφέρεστε στο αρχικό έγγραφο καταστήνων γραμμών, ε, το οποίο καταρτίστηκε το 2006, αυτό τροποποιήθηκε κατόπιν συζήτηση μεταξύ της κυρίας Δεμπαλιού και των εκπροσώπων του ΕΛΚ. Και εκπώνησαν ένα νέο εγγραφό που λέγεται ε, στις πρακτικές». Και έχουμε στο φάκελο και το έγγραφο με τις track changes ε, και εκεί βλέπετε που είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο κειμένων. Έτσι λοιπόν ε, τα μέλη του Κοινοβουλίου μπορούν να βρούμε σαφήνεια που έχουν γίνει αλλαγέ. Αλλά κανονικά θα έπρεπε να έχετε και τη δική σα ε, γλωσσική εκδοχή, γιατί λογικά έχουμε όλες τις γλώσσες διαθέσιμες. Κοιτάξτε, ένα τυπικό θέμα. Από ό,τι καταλαβαίνω, περατώσαμε τι αναφορέ που προτάθηκαν στην ομάδα Β έχουμε τα 1 9, την 1 9, 109, 102 και 61. Αυτές οι αναφορές θα μεταφερθούν στην κατηγορία Α. Συγγνώμη, αλλά καθώς μου έδωσε μια εξήγηση γραμματεία να μου πει θα έχω εγώ ένα τροποποιημένο κείμενο και στη γλώσσα μου ή όχι. Να το ξέρω θα το έχουμε και στην ε, δική μου γλώσσα ή να το μοιράσουμε στην αντιπροσωπεία. Το κείμενο με τις αλλαγές υπάρχει μόνο στα αγγλικά. Γιατί ουσιαστικά αυτό ήταν το πρωτότυπο κείμενο. Έτσι λοιπόν, το έγγραφο που έχει τις αλλαγές δεν εστάλει για μετάφραση, δεν είναι να μεταφραστεί. Zamykam nasze posiedzenie. Επομένως, ε, πέρασε τη συνεδρία. Σας ευχαριστώ.